Uh, Καλησπέρα σας. Δυστυχώς είναι ελάχιστα τα μέλη εδώ παρόντα. Έχουν στείλει βοηθούς και συμβούλους πολιτικών ομάδων, αλλά έχουν περάσει τέσσερα λεπτά από την ώρα που θα αρχίζαμε. Εν πάση Χαίρομαι που είμαστε στο σημείο 19 παρουσίαση μελέτης με ε, τίτλο ε, «Ιταλικές συμβάσεις παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων και ε, οδηγία ΤΑΔΕ». Θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες, την κυρία Μπενετάσο και την κυρία Γκομπάτο. Μοιραστείτε το χρόνο όσο θέλετε. Έχετε και παρουσίαση PowerPoint από ό,τι βλέπω. Ωραία εκατοντάδες εκατοντάδων είναι οι αναφορές σχετικά με τις παραχωρήσεις ε, ακτών και παραθαλασσιών εκτάσεων, όχι μόνο στην Ιταλία και σε άλλα κράτη-μέλη. Το θέμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο και καλωσορίζω το συνάδελφο. Τουλάχιστον είμαστε δύο. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών και τον Δόκτωρ Τζόρτζο Μούσα που μας κάλεσε να παρουσιάσουμε τη μελέτη μας ε, σε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο και είμαστε πραγματικά ε, γεμάτες τιμή. Το θέμα των ε, παραθεριστικών παραχωρήσεων και η σχετική οδηγία είναι ένα θέμα επίκαιρο και πολύ σημαντικό. Για να το παρουσιάσω σωστά, θέλω να σας παρουσιάσω κάποιες γενικές πληροφορίες πρώτα απ' όλα. Ε, για να σας εξηγήσω πρώτα απ' όλα την πολυπλοκότητα του ζητήματος αυτού. Ε, In particolare dalla complessità del να σας παρουσιάσω λοιπόν την πολυπλοκότητα του θέματος. Όπως είπα λοιπόν, το θέμα των παραθαλάσσιων παραχωρήσεων χαρακτηρίζεται από περίπλοκη νομοθεσία που αποτελεί το αντικείμενο διαφωνιών όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη. Στο Ιταλικό σύστημα, κυρίως μετά από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, για τις διάφορες Ιταλικές πρωτοβουλίες ε, ακολούθησε ουσιαστικά μια επικάλυψη πολλαπλών ε, νομοθετικών ρυθμίσεων, ξεκινώντας από ε, τον αρχικό κώδικα πλοήγησης μέχρι τον πρόσφατο νόμο εξουσιοδότησης ε, του Ιανουαρίου του 2017 που πρόβλεψε ένα σύστημα ανταγωνιστικό επιλογής του παραχωρησιούχου καταργώντας τις ανανεώσεις που χαρακτηρίζαν τον προηγούμενο νόμο στη διαδικασία αυτή θα, θα αναφερθούμε σε λίγο. Αυτή τη στιγμή ήθελα να υπογραμμίσω πως η νομοθεσία στον τομέα αυτό θέτει διάφορα ερωτηματικά. Σημαντικά, κρίσιμη σημασία είναι οι οικονομικές επιπτώσεις ε, των παραθαλάσσιων παραχωρήσεων στον τομέα του τουρισμού. Στην Ιταλία λειτουργούν περίπου 30.000 επιχειρήσεις ε, ε, και 600.000 συνολικά φορείς ε, βάσει των δεδομένων που παρέχουν οι φορείς του τομέα. Το βασικότερο πρόβλημα, δίχως άλλο, είναι αυτό της διαδικασίας επιλογής, ε, της διάρκειας της παραχώρησης, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την τοποθεσία, την αρμοδιότητα των διοικήσεων, την ποιότητα και το κόστος των παραθαλάσσιων υπηρεσιών, ε, μέχρι την ε, ελεύθερη εκμετάλλευση των παραλίων και το περίπλοκο ζήτημα του περιβάλλοντος. Δεδομένης της πολυπλοκότητας λοιπόν του νομοθετικού πλαισίου αναφοράς, μου είναι αδύνατον φυσικά εδώ να σας παρουσιάσω ολόκληρη την πολυπλοκότητα του συστήματος νομοθεσίας που υπάρχει για τέτοια θέματα στην Ιταλία. Θα περιοριστώ λοιπόν σε, ένα συνοπτικό, σε μια συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης όπως είχε πριν από τη διαδικασία παραβάση κατά της Ιταλίας το 2008 και στη συνέχεια θα περάσω στις ε, πιθανές προοπτικές μεταρρύθμισης ε, εν ώψη της σημαντικής απόφασης ε, του, δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 14 Ιουλίου του 2016 που φαίνεται να επιβάλλει όπως βλέπουμε μια αναθεώρηση ε, της ε, σημερινής νομοθεσίας η οποία δεν μπορεί πλέον να αναβληθεί. Όσον αφορά το σύστημα που καθορίζει ο δικός μας Ιταλικός Κώδικας Πλοήγησης χαρακτηρίζεται από ε, ένα νομοθετικό πλαίσιο που ονομάζεται το, έτσι όπως το ονομάζουμε εμείς, δίκαιο, δίκαιο επιμονής, δηλαδή το δικαίωμα του ε, εξερχόμενου ε, παραχωρησιούχου να αποτελέσει το αντικείμενο προτι... Ε, να έχει προτιμησιακό προνόμιο σε σχέση με τους υπόλοιπους όπως προκύπτει μετά από την διαδικασία παραβάσης κατά της Ιταλίας του 2008. Δεδομένου αυτού του συστήματος που περιγράφεται στον κώδικα ε, ναυσιπλοείας που χαρακτηρίζεται από μεγάλο κατακαιρματισμό, η επόμενη νομοθεσία απογοήτευσε και κατάργησε ουσιαστικά τις ε, αρχές ε, που είχαν εμπνεύσει την αρχική νομοθεσία. Έτσι εισήχθη μια μέγιστη διάρκεια για τις παραχωρήσεις 20 ε, ετής όπως ορίστηκε τελευταία από το νόμο 296 του 2006 που τέθηκε σε το 2007 και μειώθηκε η διακριτική ευκαιρία της διοίκησης. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ανάκληση. Ωστόσο, η πιο σημαντική παρέμβαση ήταν με τη διαδικασία επιπαραβάση που υπέστη η Ιταλία το 2008. Μια διαδικασία επιπαραβάση που, ωστόσο, πρέπει να πούμε, είχε προ, προ, προηγηθεί αυτής μια επισήμανση από τη δική μας την Ιταλική Αρχή Αντιτράστα, την Αρχή ε, Διασφάλισης του ε, Ανταγωνισμού από τον Οκτώβριο του 2008 και από ε, μία απόφαση του δικού μας Βουλίου της Επικρατείας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Αγοράς είχε ζητήσει να ανοιχτεί ο τομέας όπως ήταν απαραίτητο ώστε να χρησιμοποιηθεί ένας ε, κανόνας ε, διαδικαστικός ε, για να, είναι, να έχει δημόσια προβολή η εκχώρηση των αδειών. Με την απόφαση της 7ης Δεκεμβρίου του 2000, όπως ξέρουμε, είχε επιβληθεί η γενικότερη ισχύ τη αρχή τη διαφάνεια και για τι συμβάσει που συνάπτονταν στο πλαίσιο τη εφαρμογή συγκεκριμένων οδηγιών κοινοτικών. Στη δική μα περίπτωση λοιπόν και για τι παραχωρήσει αγαθών που όπω γνωρίζουμε εξαιρούνται από τον τομέα εφαρμογή ε, τη οδηγία 23 του 2014 όπω προκύπτει ρητά από την 15η αιτιολογική σκέψη της ίδιας ε, αυτής ε, οδηγία και όπως επικυρώνεται πιο πρόσφατα από την ίδια απόφαση του δικαστηρίου in present δεν θέλω να ασχοληθώ με την διαδικασία παραβάση εδώ, ούτε θεωρώ απαραίτητο το να επανέλθουμε στα ε, προδικαστικά ζητήματα που τέθηκαν σε σχέση με αυτό την Ιταλική νομοθεσία που οδήγησε σε ε, παράταση των παραχωρήσεων ε, μέχρι το 2020 μέχρι να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό θα μιλήσει η συνάδελφος Αραγκομπάτο. Θα περιοριστώ στο να υπενθυμίσω ότι η απόφαση του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, περιλαμβάνει όπως το βλέπω εγώ, ε, χρήσιμες διευκρινήσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Volkenstein ε, που μπορούν να αποτελέσουν σημεία αναφορά και για τον Ιταλό νομοθέτη εν ώψη της ε, πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση του τομέα. Πράγματι, το δικαστήριο, παρότι διαπιστώνει ότι γενικά η οδηγία Βολκενστάιν βασίζεται σε μια εσωτερική νομοθεσία που προβλέπει ε, παρατάσεις των σημερινών παραχωρήσεων αυτόματα, χωρίς διαδικασία επιλογής, Επιβεβαιώνει όμως επίσης ότι οι επιμέρους εθνικές αρχές μπορούν να υιοθετήσουν λύσεις βασισμένες ε, σε εύλογη ε, εμπιστοσύνη ώστε να ε, χρησιμοποιηθούν άλλοι, άλλοι όροι ως άλλοι παράγοντες ως ε, σημεία αναφορά. Θα το δούμε αυτό στην παρέμβαση τη Αραγκομπάτο. Πρέπει να πούμε ότι το ζήτημα των παραθαλάσσιων παραχωρήσεων στη δική μα μελέτη δεν εξετάστηκε μόνο βάσει του εσωτερικού δικαίου, του Ιταλικού δικαίου, αλλά και συγκριτικά με αναφορά στα διαχειριστικά ε, συστήματα που χρησιμοποιούν άλλα κράτη-μέλη ώστε να επαληθευτεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του Ιταλικού συστήματος σε σχέση με άλλα συστήματα νομοθετικά. Πράγματι, εξετάσαμε τις εμπειρίες στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Κροατία και στην Ελλάδα. που θεωρούνται κατά κάποιο τρόπο ανταγωνιστές της Ιταλίας διότι από άψη γεωγραφική, γεωγραφικής μορφολογίας έχουν τεράστια ακτογραμμή οι μέσες θερμοκρασίες ε, εποχιακά είναι ίδιες με τις Ιταλικές και επίσης και όσον αφορά τις ε, διοικήσεις ε, στα κράτη-μέλη. Αυτά υπάρχει η ίδια κατανομή αρμοδιοτήτων και λειτουργούν πολλά επίπεδα διακυβέρνηση όπως και στην Ιταλία. Παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε ορισμένες κοινέ τάσεις. Πώς δηλαδή μεταξύ των διαφόρων διοικητικών συστημάτων υπάρχουν σημαντικές ε, συγκλήσει. Σε σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη παρατηρείται μεγάλη προσοχή στα ολοκληρωμένα ε, προφίλ διαχείρισης ε, των παραθαλάσσιων περιοχών για την προστασία των αγαθών αυτών και των στοιχείων τους. Αυτή η προσοχή σε περιβαλλοντικά θέματα είναι σαφής κυρίως στη Γαλλία που συχνά αναφέρεται ως μοντέλο ε, διαχείρισης ε, των παραθαλάσσιων αγαθών, διότι το γαλλικό σύστημα φαίνεται να προσανατολίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ε, περιβαλλοντική προστασία των θαλάσσιων αγαθών. Επίσης ευνοεί τη γενική χρήση από, το, από τον πληθυσμό περισσότερο από ό,τι επιχειρήσεις. Αυτό το βρίσκουμε στο Μπιμπιόνο Σαμικέλε στην Ιταλία που θα εμβαθύνουμε αργότερα. Ήθελα να πω ότι αυτή η εστίαση στα περιβαλλοντικά θέματα υπήρχε και στο δικό μας κώδικα ναυσιπλοείας, ειδικότερα στο άρθρο 37, δεύτερη παράγραφος πρώτο εδάφιο, που είναι η διάταξη που αφορά την υποχρέωση του παραχωρησιούχου να, να, αφαιρεί όλα τα ε, κινητά ε, ε, αντικείμενα στο τέλος της παραθυριστικής περίοδου ώστε να προστατευθεί η παραθαλάσσια περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο αλλά υπάρχει και άλλος ένας δεύτερος στόχος που προκύπτει από την ανάλυση δηλαδή η ανάγκη βελτίωσης της διαχείρισης των ε, αγαθών των στοιχείων του αγιαλού ε, που σε πολλά κράτη-μέλη φαίνεται να πραγματοποιείται μέσω μηχανισμών επιλογής, διαδικασιών, διαφάνειας για την επιλογή του παραχωρησιούχου. Μπορεί κανείς να πει ότι όλο και συχνότερα και σε περιφερειακό επίπεδο παρατηρείται αυτή η μεγαλύτερη προσοχή μέσω των ε, ε, δημόσιων διαδικασιών. Όσον αφορά την Ιταλία, η αξία των αρχών της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, της ίσης μεταχείρισης αφορά και εκτιμένο στην Ιταλική ε, νομολογία βάσει των αποφάσεων που, είπα, που ανέφερα προηγουμένω του Συμβουλίου τη Επικρατείας αλλά και των αρχών ανταγωνισμού και αγοράς. Προκύπτει και κάτι καινούριο που έχει κυρωθεί πλέον και σε νομοθετικό επίπεδο. Ε, αναφέρομαι στην μεταρρύθμιση που αφορά τη μεταβίβαση αγαθών από το κεντρικό κράτος στις ε, περιφερειακές, στις τοπικές αρχές. Παραμένει ωστόσο ένα πρόβλημα, ένα βασικό πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τον Ιταλό νομοθέτη στο μέλλον, όχι μόνο τον Ιταλό. Θα πρέπει να εντοπιστεί μια συγκεκριμένη διαδικασία παραχώρησης η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει αφενός τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προκύπτουν από το ενωσιακό δίκαιο, αφετέρου τις απαιτήσει προστασίας ε, του εξερχόμενου παραχωρησιούχου. Μια πτυχή που σχετίζεται στενά μάλιστα με τη διάρκεια της παραχώρησης η οποία από αυτή την άποψη θα πρέπει και αυτή να αναθεωρηθεί διότι και εδώ έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Στη Γαλλία η μέγιστη διάρκεια που προβλέπεται είναι 12 έτη για τις παραθαλάσσιες παραχωρήσεις. Στην Ιταλία είναι 20 βάσει της σημερινής νομοθεσία, Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, για παράδειγμα, είναι δυνατόν να φτάσει κανείς και στα 75 έτη για τις ε, δομές ε, ε, μεγαλύτερου οικονομικού βάρους. Και στην Κροατία, όπου ισχύει αυτός ο ο κανόνας του δημόσιου διαγωνισμού υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου είναι δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη διάρκεια της παραχώρησης. Αντιθέτως όσον αφορά τη διαχείριση του αγαθού ε, συνοδεύονται από παρεμβάσεις αναδόμησης των ε, παραθαλάσσιων περιοχών. Πώς να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Η διέξοδος, ε, κατά την άποψή μου, θα εστιάζεται στις πληροφορίες που έρχονται από το δικαστήριο, ε, θα βασιστεί σε στενή συνεργασία και διάλογο μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επιμέρους ιταλικών και εθνικών αρχών, διότι η οδηγία Βόλκενσταιν εξηγεί ε, πώς μπορούμε να βρούμε ομογενείς λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποφεύγοντας ε, την επιβολή υπερβολικών περιορισμών Εν συντομία, ποιες είναι οι πιθανές παρεμβάσεις. Πρώτον, είναι απαραίτητο να γίνει ένας γενικός συντονισμένος προγραμματισμός ε, των παραλίων και των αγιαλών, των παραθαλάσσιων περιοχών, διότι η διαχείριση αυτή η χωροταξία χρειάζεται ε, ε, πληροφορίες πιο σαφείς και διαφανείς. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ενίσχυσης του συστήματος πληροφοριών των παραθαλάσσιων περιοχών που υπάρχει στην Ιταλία από το 1993 να υπάρχει δηλαδή μια βάση πληροφοριών για το πλήθος και τη σύνθεση των ε, τοποθεσιών, διότι έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να έχουμε μια εναλλακτική νομοθεσία από την υπάρχουσα, όπως διευκρινίζει το δικαστήριο που επιβεβαίωσε σαφώς ότι ε, μια εναλλακτική νομοθεσία θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη μια δέσμευση που θα σχετίζεται με την με τον ε, σπανίου χαρακτήρα των πόρων ε, και των υπηρεσιών αυτών. Ε, αν θέλετε αργότερα, επειδή είναι πολλά τα θέματα και πληροφορίες, θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε. Ή να δούμε τι, ποιες είναι οι πιθανές μελλοντικές νομοθεσίες και ποιες είναι οι δυνατές πρόπτικες που έχουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Είναι το τμήμα μελετών C, το Policy Department, στο οποίο αναθέσαμε τη μελέτη αυτή και το έπραξαν και με έναν τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικό όσο και χρήσιμο. Λοιπόν, η μελέτη αυτή ε, ε, θα διαβαστεί και θα δοθεί και συνέχεια, όχι μόνο από τα μέλη της Επιτροπής μας, αλλά από όλους τους Ευρωβουλευτές. Είναι προς όφελος όλων των Ευρωβουλευτών. Εσείς μακρηγορήσατε. Ε, παρακαλώ, κυρία Γκομπά, το σύντομα να συμπληρώσετε μόνο. Πολύ λίγα λεπτά. Μόνο τρία λεπτά θα χρειαστώ για να σας ε, παρουσιάσω κάποια σημαντικά σημεία τα οποία ανέδειξε η μελέτη μας ε, βάσει της ανάλυσης ε, της διαδικασίας σε παραβάση που έκλεισε ενώπιν της Ιταλίας το 2010 και της προδικαστικής απόφασης του 2016. Αυτά τα σημεία μπορούν να συνοψιστούν σε πέντε διαπιστώσεις νομικές που επειδή έχουν παρασχεθεί από του θεσμού των ευρωπαϊκών οργάνων ισχύουν ομοιόμορφα για όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση. Εν συντομία λοιπόν, πρώτον, πρώτο, ε, εθνικές διατάξεις που επιτρέπουν οριζόντια μέτρα που εφαρμόζονται απευθείας σε όλους τους παραχωρησιούχους αλλά αυτά δεν συμβαδίζουν με το άρθρο 49 της συνθήκης και το άρθρο 12 της οδηγίας. Δεύτερο σημείο αφορά τις εθνικές αρχές οι οποίες πρέπει να αξιολογούν αν οι παραχωρήσεις εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 12 της οδηγίας ή στο άρθρο 49 της συνθήκης. Στην πρώτη περίπτωση, όπως μας τόνισε ε, το δικαστήριο, οι παραθαλάσσιες παραχωρήσεις εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 12 εάν αφορούν σπάνιους φυσικούς πόρους. Στη δεύτερη περίπτωση, αν λοιπόν εκεί δεν ισχύει, αν δεν εντάσσονται στο άρθρο 12, οι εθνικές αρχές ε, έχουν την αρμοδιότητα να επαληθεύσουν κατά πόσο οι παραχωρήσεις παρουσιάζουν διασυνοριακό ε, ενδιαφέρον, βέβαιο και συνεπώς εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49. Τρίτο σταθερό σημείο σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις είτε ισχύει το άρθρο 12 της οδηγίας είτε ισχύει το άρθρο 49 της συνθήκης η παραχώρηση κρατικής περιουσίας πρέπει να πραγματοποιείται βάσει διαδικασιών επιλογής των πιθανών ε, υποψηφίων, διαφανών και μη διακριτικών. Τέταρτο σημείο, στην ε, σύνταξη των διαδικαστικών κανόνων για τη διαδικασία επιλογής οι εθνικές αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη επιβεβλημένα κίνητρα ε, κοινού συμφέροντος που πρέπει να συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης. Ε, τέτοια επιβεβλημένα κίνητρα μπορούν να είναι στόχοι κοινωνικής πολιτικής και προστασία του περιβάλλοντος πέμπτο και τελευταίο σταθερό σημείο και με αυτό θα κλείσω. Δυνάμει των Γενικών Αρχών του Ενωσιακού Δικαίου περί ε, εύλογης ε, παραχώρησης οι εθνικές αρχές πρέπει κατά περίπτωση να αξιολογούν τη θέση των εξερχόμενων παραχωρησιούχων. Η αρχή της εύλογης παραχώρησης επιτρέπει οι επενδύσεις των εξερχόμενων ε, παραχωρησιούχων να παραμένουν καθώς έχει ληφθεί υπόψη η παράταση των ε, ε, παραχωρήσεων. I thank you very much and... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρειάζεται εκβάθρον ανανέωση η νομοθεσία για τις παραλίες και τον Αγγελό στην Ιταλία. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία και οι πρόσφατες αποφάσεις δικαστικές και τα συμπαρομαρτούντα θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και σε μεγάλο βάθος. Δεν είναι του παρόντος τώρα να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αλλά παρακαλώ να διαβάσετε όλη τη μελέτη. Διατίθεται εδώ στην είσοδο της αίθουσης και μπορείτε να τη βρείτε. Τώρα, ο κύριος Λεκορντάρη ε, απουσιάζει, εξ όσων κατάλαβα, Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιος είναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yes, thank you for giving me the... Ευχαριστώ πολύ. Οι υπηρεσίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελαν καταρχήν να ευχαριστήσουν την Επιτροπή σας που μας καλέσατε σε αυτή τη συνάντηση και πρέπει να σας πω πως καταγράφουμε τα όσα έχετε στη μελέτη, τα στοιχεία, τα δεδομένα, και την ανάλυση αυτών που κάνετε. Επίσης καταγράφουμε ιδιαίτερα πως το ΔΕΚ έχει προσφέρει διευκρινήσεις που είναι πολύ σημαντικές για το που εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι διευκρινήσεις αυτές θα πρέπει οπωσδήποτε να κατευθύνουν όλες τις εθνικές αρχές σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να ανταποκριθούν όπως πρέπει στις αρμοδιότητες που έχουν για διαχείριση της γελίου ζώνης ε, και βέβαια πάντα σε περίπτωση δικαστικών διενέξεων. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα ξεκάθαρο εθνικό νομικό πλαίσιο σύμφωνα με τα όσα έχει αποφασίσει το ΔΕΚ έτσι ώστε να εξασφαλίσει τη νομική βεβαιότητα. Και αυτό πάντα είναι ευπρόσδεκτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την εφαρμογή αυτών των αρχών σε όλη την επικράτεια, επαναλαμβάνω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επαναλαμβάνω, συνεχίζουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Thank you. Thank you very much. Well, this is now a moment. Πολύ ωραία. Φτάσαμε λοιπόν την στιγμή ε, που δεν θα συζητήσουμε πλέον τις μεμονωμένες αναφορές, το έχουμε αποφασίσει προηγουμένως, αλλά για τις ε, παραχωρήσεις ε, παράκτιων ζωνών, εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, αν έχετε κάποιες διευκρινήσεις που θέλετε για τη μελέτη, νομίζω ότι μπορώ να σας δώσω το λόγο. Ο κύριος... Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις προς τις ε, δύο προσκεκλημένες. Η πρώτη να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε η πρώτη μελήτρια, ε, υπήρξε τρόπος να δείτε το, έχετε δει το τελευταίο Ιταλικό νομοσχέδιο. Σχετίζεται αυτό με τα απορίσματα της μελέτης σας και συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς νόμους. Υπάρχει κάποια αντιστοιχεία και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω πώς ερμηνεύεται την έννοια των περιορισμένων Ισπάνιων φυσικών πόρων γιατί και από αυτού έχουν γίνει πολλές συζητήσεις γιατί περιορισμένη είναι μία έννοια, Ισπάνιες είναι άλλη έννοια. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω στην πρώτη ε, ερώτηση και θα δώσω τη συναδελφό μου στην δικηγόρο, στην νομική Γκομπάτο για τη δεύτερη ερώτηση. Το νομοσχέδιο αυτό ήθελα να το αναφέρω διότι έχουμε ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι φαίνεται να υιοθετούνται κάποιες από τις υποδείξεις του δικαστηρίου σε αυτό το νομοσχέδιο της 27ης Ιανουαρίου του 2017. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, το νομοσχέδιο αυτό εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο. Δυστυχώς αναβλήθηκε η εξέταση στη Γερουσία ε, καθώς λύθηκαν ε, τα νομοθετικά σώματα γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο στην Ιταλία οπότε 28 Δεκεμβρίου έλυσε τα κοινοβουλευτικά σώματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οπότε δεν προλάβαμε να γίνει εξέταση και στο Ιερουσία. Όσον αφορά εμάς από όσο είδαμε και αναλύσαμε ως Πανεπιστήμιο της Πάδοβας και σε, μια πρόσφατη, σε ένα πρόσφατο συνέδριο που έγινε τον περασμένο Μάιο για το θέμα αυτό πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο κατά την άποψή μα περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία θετικά τα οποία κινούνται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. Κυρίως διότι υιοθετεί επακριβώς την αρχή της, του ανταγωνισμού ε, όπως αναγνωρίζεται από τη δική μας εσωτερική νομολογία και διοικητική αλλά και συνταγματική αλλά και από την εγκυητική αρχή. Το σταθερό σημείο είναι οι διαδικασίες διαφάνειας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο διότι υιοθετεί και τις υποδείξεις του δικαστηρίου όσον αφορά την ευλογική εμπιστοσύνη. Βασίζεται, λοιπόν, θέτει διάφορα κριτήρια ε, ε, μεταξύ λοιπόν των αρχών και των κριτήριων που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσανατολισμό ε, περιλαμβάνεται το ολοκληρωμένο, η ολοκληρωμένη άποψη του κόστους ε, που έχουμε δει και στη Γαλλία και στην Κροατία σε πιο πρόσφατη νομοθεσία. Θέτει λοιπόν αυτή την αρχή της θεμητής εμπιστοσύνης μεταξύ των βασικών αρχών, υπενθυμίζοντας και το ε, άρθρο 12.3 της οδηγίας Βολκενστάιν, θέτει και το ζήτημα της κεκτηθήσας επαγγελματικότητας για τον νέο παραχωρησιούχο σε περίπτωση διαγωνισμού. Από ό,τι φαίνεται όμως ε, βάζει ένα σύστημα δύο ταχυτήτων σε σχέση με αυτό που υπάρχει στη Γαλλία ή και στην Κροατία. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη αυτό, ε, η ε, δέσμευση, που σχετίζεται με το σπάνιο χαρακτήρα αυτή τη εξήγηση Άρα λαμβάνει δηλαδή υπόψη, προβλέπει μία περίοδο μεταβατική των παρατάσεων όπου θα πρέπει να ορίζεται μια παράταση ώστε να μπορέσει ο ιστορικός κανονισμό να προσαρμοστεί φυσικά περιορισμένη παράταση αλλά επ' αυτού η συζήτηση ήταν πολύ μεγάλη. Δεν έχει καταφέρει να επιτευχθεί συμφωνία γι' αυτό. Η μεταβατική αυτή περίοδος που θα συνοδεύεται από κάποια δημόσια στοιχεία για τις μη εκχωρημένες παραλίες ταυτόχρονα όπως το καταλάβαμε εμείς στην Πάδοβα, φαίνεται να υιοθετείται μια διαφοροποιημένη ε, προσέγγιση όσον αφορά τις προηγούμενες παραχωρήσεις ε, που λήγουν. Ε, σε αυτή την περίπτωση, κατά την άποψή μου, δεδομένης της εφαρμογής των μηχανισμών δημοσιοποίησης για θέματα ανταγωνισμού και μέσω και της χρήσης της δημόσιας διαβούλευσης, όπως η Enquête Publique στη Γαλλία, θα μπορούσε να προβληθεί αυτού του είδους δηλαδή δημοσιοποίηση για μηνές παραχωρήσεις ταυτόχρονα δημιουργεί και ένα δίκτυο προστασίας για τους σημερινούς επιχειρηματίες όχι μόνο όπως είπαμε μέσω του καθορισμού της, περίοδου, της μεταβατικής περίοδου αλλά εισάγοντα και διατάξεις που προβλέπουν ε, την ε, θεμητή εμπιστοσύνη και έτσι βλέπω στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, λαμβάνεται υπόψη, λαμβάνεται υπόψη τα αιτήματα που αφορούν ε, την βιωσιμότητα, την περιβαλλοντική, αλλά και τη βελτίωση των ε, συνθήκων ε, στις παραλίες. Οπότε ουσιαστικά ζητήματα περιβάλλοντος, ανταγωνισμού και θεμητής εμπιστοσύνης λαμβάνεται υπόψη το νομοσχέδιο αυτό το οποίο θα πρέπει φυσικά να επανεξεταστεί, να βελτιστοποιηθεί όσον αφορά τις διάφορες ε, αρχές αυτές, αλλά σίγουρα είναι ένα καλό ε, κείμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία, θεωρούμε εμείς. Ε, θεωρητικά δηλαδή συμφωνούμε εμείς. Το συζητήσαμε και σε ένα συνέδριο και συμφωνήσαμε όλοι για αυτά τα σημεία. Ευχαριστώ. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση που αφορά την εφαρμογή του αρθρού 12 αδειοδοτήσεις περιορισμένες εδώ θα ήθελα να αναφορθώ για να σας απαντήσω στη θέση που υιοθέτησε ο εισαγγελέα στην ε, υπόθεση Προμομπρέζα Εμέλης στα σημεία 70 και 72 των συμπερασμάτων του εισαγγελέα. Τι λέει το δικαστήριο μέσω του εισαγγελέα. Λέει ότι όπως εσείς αναφέρατε στην ερώτησή σας, το άρθρο 12 εφαρμόζεται σε παραχωρήσεις περιορισμένους διότι σχετίζονται με σπάνιους φυσικούς πόρους. Ο εισαγγελέα ανέφερε ότι τέτοιου είδου ε, παραχωρήσει θαλασσιών περιοχών, παραθαλάσσιων περιοχών ε, παραχωρούνται από Ιταλικού ε, νόμους. Σχετίζονται με γεωγραφικού χώρου περιορισμένους. Βάσει αυτού, λέει ο εισαγγελέα, θεωρείται ότι υπό αυτές τις συνθήκες εφαρμόζεται το άρθρο 12 στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, λόγω του δημοτικού χαρακτήρα των αρχών που παρέχουν αυτές τις άδειες. Thank you very much and I'm sure that... Ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε λόγο να επανέλθουμε και να αποτανθούμε ξανά σε εσά όταν θα λάβουμε και είμαι βέβαιη ότι θα λάβουμε περισσότερες αναφορές για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και καλή τύχη και καλή συνέχεια στις μελλοντικές σας εργασίες για αυτό το τόσο σημαντικό ε, θέμα για την Ευρώπη. Ευχαριστώ και πάλι. Προχωρούμε, συνάδελφοι, στο επόμενο θέμα στη μέρη διάταξη. 20. Αναφορά 336 του 2012, 721 του 2014 και 1141 επίσης του 2014 για τη συστηματική κοπή της ουράς των χειριδίων στη Δανία και στη Σουηδία και στη Μεγάλη Βρετανία. Ξαφνικά ε, γεμίσαμε Σκανδιναβούς εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στην Ιωάννα Σπάβε που είναι εδώ όχι για πρώτη φορά και νομίζω ότι έχετε και εσείς ένα PowerPoint το πολύ πέντε λεπτά παρακαλώ, αλλά όπως γνωρίζετε ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Humane Society International και των συναδέλφων ε, αναφερομένων ε, για ε, τα θέματα της καλής ε, κτηνοτροφίας. Αυτή η σημαντική κοπή της ουράς των χείρων είναι 15 χρόνια παράνομη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 2003. Ωστόσο, το 90% των χείρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να έχουν κομμένη την ουρά. Αυτό το έχει τονίσει και η Κόπα Κοζέκα και υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο νόμος είναι πολύ καλά γραμμένος, δεν ε, απαγορεύει κάθε κοπίουρας, αλλά θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσουν οι χειροτρόφοι ε, να βελτιώσουν ε, τη διαβίωση των χειριδίων για να μην έχουμε τέτοιο κανιβαλισμό που δαγκώνουν την ουρά τους. αν γίνεται κάτι τέτοιο, να κοπεί ουρά, αλλά και πάλι από εκεί και πέρα να βελτιωθούν οι συνθήκες εκτροφής για να σταματήσει αυτός ο καρεβαλισμός στη Σουηδία και τη Φιλανδία έχει απαγορευτεί πλήρως αυτή η πρακτική στη χειροτροφία. Οι συνάδελφοι του Compassion in World Farming έκαναν έρευνες και έδειξαν ότι περισσότεροι χειροτρόφοι δεν κάνουν καμιά σοβαρή προσπάθεια να βελτιώσουν τις συνθήκες εκτροφής και κατά ε, σύστημα κόβουν τις ουρές. Χρειάζονται ε, κάποια εμπλουτιστικά υλικά, παιχνίδια ουσιαστικά και οι χείροι για να μην ε, δαγκώνουν την ουρά των άλλων χειριδίων. Ε, δηλαδή θα πρέπει να έχουν άχυρο ή ξύλο γιατί είναι περίεργα ζώα και θέλουν κάτι για να απασχολούνται. Οι περισσότεροι χειροτρόφοι τι κάνουν, δίνουν πλαστικά παιχνίδια ή μεταλλικές αλυσίδες. Ακόμα και μετά που η ΕΦΣΑ ή ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισαν ότι δεν βοηθούν τέτοια υλικά. 63% των χειροτρόφων δίνουν απλώς κάποιες μεταλλικές αλυσίδες για να παίζουν τα γουρούνια ή ε, πλαστικά παιχνίδια που δεν τους ενδιαφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια πιέζει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την οδηγία σωστά. Το 2016 εξέδωσαν ε, συστάσει για τις δράσεις που πρέπει να γίνουν για να περιοριστεί η κοπή της ουράς και ο κανιβαλισμός μεταξύ χειριδίων. Ε, το 2017, πέρσι δηλαδή μόλις, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κάποια ενημερωτικά δελτία σχετικά. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη τα περισσότερα δεν κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να περιορίζουν τη συστηματική κοπή της ουράς και να δίνουν εναλλακτικέ λύσεις στους χειροτρόφους. Το 2018 θέλουμε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να φροντίσει να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία και με ποιες προθεσμίες όταν τα κράτη-μέλη δεν δίνουν λεπτομερή προγράμματα ε, δράσης ε, με γρήγορη και ουσιαστική συμμόρφωση. Σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσφεύγει επί παραλήψη. Δεν μπορεί αυτή η υψηλή έλλειψη συμμόρφωσης να γίνει ανεκτή στο μέλλον. Ζητούμε επιμόνως από την Επιτροπή σας ε, να διατηρήσει ανοιχτή την συμπεριφορά και να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα κράτη-μέλη δεν συμμορφώνονται σωστά με την νομοθεσία και δεν απαγορεύουν τη συστηματική κοπή τη ουράς των χειριδίων. Και δεν δίνουν ε, στα γουρούνα και αυτά τα υλικά που χρειάζονται για να του αποσπάσουν την προσοχή από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δίνω το λόγο λοιπόν κατευθείαν στο Φέντερικ ε, Φέντερλε, ο οποίος όταν υπευλήθη αναφορά δεν ήταν ευρωβουλευτής, αλλά είχε υποβάλει αναφορά στην Επιτροπή μας. Ήταν ένα δείγμα εμπιστοσύνης. Πριν σας δώσω το λόγο λοιπόν, θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα έχει κάνει η Επιτροπή μας και νομίζω ότι θα πρέπει να το έχω κάνει ε, ξεκινώντας την παρουσίαση. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και έχουμε επενδύσει πολλή προσπάθεια εδώ και κάποιες από τις δράσεις που αναλάβαμε ήταν η μελέτη που ζητήσαμε το 2014, οι επιστολές που στείλαμε στον κύριο Κάιτη στον Επίτροπο, για μια ενδεχόμενη διαδικασία παραβάση. Θα επανέλθω επίσης τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Άγκρη, ε, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα, όπως επίσης και στην ΕΝΒΗ η οποία δεν μας απάντησε Οπότε πρέπει να σας πω πως έχουμε πραγματικά αναλάβει δράση. Και Φρέντρικ λέγοντας αυτά σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για το γεγονός που κρατήσατε το φάκελο αυτό ανοιχτό γιατί πιστεύω ότι η Επιτροπή Αναφορών αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι όταν ασχολείται με τέτοιου είδους ε, φακέλους. Για να συμπληρώσω τα όσα ακούσαμε, ξέρουμε πως το ο κανονισμός έδωσε 10 χρόνια στα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν. Άρα λοιπόν το 2013 έπρεπε να έχουμε πλήρη συμμόρφωση. Το 2008 το Συμβούλιο έθεσε μια σειρά κανόνες για το πώς μπορεί κανείς να συμμορφωθεί με την ε, διαδικασία, με τον κανονισμό για τους χείρους και πρέπει να σας πω πως έχουν περάσει τόσα χρόνια και πάλι δεν έγινε. Παρόλο που έχει προσπαθήσει να προωθήσει το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια ε, στεναρή ψηφοφορία στο Στρασβούργο, η Επιτροπή Αναφορών, Προεδρία και η Επιτροπή Ένβη και η Επιτροπή Άγκρη και όλα αυτά. Τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερα προσφυλή ε, και ανησυχούν ιδιαίτερα θα έλεγα τον Ευρωπαίο πολίτη. Στην τελευταία μεγάλη έρευνα που έγινε το Φεβρουάριο πέρυσι, ο Επίτροπος κ. Αντρουκάητη είπε πως υπάρχει ε, ισχυρή στήριξη έτσι ώστε να αλλάξουν κάπως τα πράγματα ε, σε επίπεδο κρατών μελών και νομίζω ότι με τα σχέδια δράσης τα οποία είναι ε, αρμόδια να παρουσιάσουν τα κράτη-μέλη κάτι θα γίνει. Επίσης η βασική ιδέα που θα πρέπει να δούμε είναι το πώς μεταχειριζόμαστε τα ζώα. Γιατί όταν χρειάζεται κανείς να κόψει ε, ε, την ουρά από τα χειρίδια είναι γιατί η κτηνοτροφία γίνεται σε κακές συνθήκες. Εάν ε, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες απασχόλησης των χειριδίων και υπαρκής χώρος δεν θα δαγκώνουν το ένα την ουρά του άλλου. Οπότε δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε κοπή της ουράς αυτές. Γίνεται καμιά φορά για ιατρικούς λόγους. Αλλά βλέπετε πως πολλά κρατημέλη διαφορούν για το θέμα. Ξέρω πως ο συνάδελφος, ο οποίος είναι πρόεδρος είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευζοία των Χείρων. Ε, θα λάβει το λόγο μετά από μένα, αλλά νομίζω ότι η Δανία ε, πρέπει να σας πω πως ε, είναι πολλοί γεωργοί στη Δανία που δεν κόβουν τις ουρές από τα χωρίδια. Ξέρετε πως στη Σουηδία έχουμε καλές τιμές, καλή παραγωγή και δεν έχουμε και Οπότε είναι απλώς οι άθλιε συνθήκε διαβίωσης που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν αυτή την τακτική. Οπότε ελπίζω να κρατήσουμε το θέμα ανοιχτό, την αναφορά αυτή ανοιχτή πριν, ε, και να μην την κλείσουμε πριν δούμε τα σχέδια δράσης των κρατών μελών. Και ευχαριστώ του συναδέλφου που ενδιαφέρονται, που πιέζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο γιατί τελικά έχει να κάνει με του εκπροσώπου των κρατών μελών οι οποίοι ωραία λόγια λένε στη συναντήσει του Συμβουλίου και παρουσιάζουν στεναρές ε, θέσει τι οποίε μετά δεν εφαρμόζουν και τελικά τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε και του κανόνε του οποίου έχουμε θεσπίσει εμεί οι ίδιοι άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλή ερώτηση που κάνετε. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μαγκύρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στη σημερινή συνεδρίαση. Πιστεύω πως η παρουσίαση ε, από το ΣΟΑΜ ήταν πολύ καλή και θα συμπληρώσω τα όσα είπε η συνάδελφος για να δείτε ποια είναι η δράση που έχουμε αναλάβει. Έχουμε γράψει επιστολές στα κράτη-μέλη να δούμε τι γίνεται με τα εθνικά σχέδια δράσης και είναι ο τέλη Ιανουαρίου 2018 η καταληκτική προθεσμία για την κατάθεση των σχεδίων αυτών. Θα τα εξετάσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και έχουμε στείλει και κάποια εγχειρίδια και εκπαιδευτικά κείμενα στην, ε, στο σχετικό κλάδο ε, και κάναμε συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους, με ε, τον κλάδο, τη εκτροφή, του ενημερώσαμε. Αυτά λοιπόν και ανάλογα και με τα σχέδια δράσης, αν χρειαστεί θα αναλάβουμε δράση για να είμαστε σίγουροι πως θα αποφεύγεται ε, το πρόβλημα του δαγκώματος της ουράς ε, μεταξύ χειριδίων και κατ' επέκταση να αποφεύγουμε και την κοπή της ουράς. Ποιος ευρωβουλευτής θέλει το λόγο. κυρία Άουκεν. Ναι, ευχαριστώ. Θα μιλήσω για αλλαγή διδανικά. Πραγματικά είναι μια περίπτωση που αφορά πάρα πολύ και τη Δανία και ξέρω όσοι παρακολουθούν τη συζήτηση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη Δανία είναι πολύ ε, το 2014 από τι ευρωεκλογέ είχε συγκεντρώσει επίση την προσοχή του κόσμου αυτό το θέμα και τότε μας αποσχολούσε ε, από τη σκοπιά της τρέβλου του ανταγωνισμού ε, απέναντι στη Σουηδία και κάποιες άλλες χώρες, λίγες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σέβονται την οδηγία και την ομοθεσία. Δεδομένου ότι η μεγάλη ε, πλειονότητα των κρατών μελών δεν συμμορφώνεται. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί Θα επιβληθούν τώρα κυρώσεις για τις χώρες που δεν συμμορφώνονται. Μέχρι τώρα συνέχιζαν την πρακτική του παρελθόντος ε, χωρίς καμία αλλαγή. Ακούμε ακόμα χειροτρόφους στη Δανία να λέγουν ότι η ε, βιαιότητα και το απάνθρωπο για τα ζώα είναι να μην τους κόβει στην ουρά ακριβώς τα χειρίδια. Ε, και στα χειροστάσια η κατάσταση είναι τόσο εκτρή που ε, ε, τα, τα χειρίδια δαγκώνουν το ένα την ώρα του άλλου. Ελπίζω κάτι να γίνει και να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στα κράτη-μέλη. Εμείς έχουμε υπουργό που συνήθως είναι 100% στην πλευρά των χειροτρόφων. Αλλά υπάρχει και ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος που είναι μια περίεργη δανέζικη κατασκευή, ο οποίο βγήκε και είπε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη συστηματική κοπή τη ουράς των χείρων. Εγώ δεν έχω την παραμικρή ε, υποψία, η ένδειξη ότι το εννοεί αυτό που λέει. Ας ελπίσουμε ότι το εννοεί. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πιέσει τα κράτη-μέλη να σέβονται τις υποχρεώσεις τους και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να συμμορφώνονται προς αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αδρανήσει λίγο μέχρι σήμερα σε αυτό το τομέα και θα ήθελα να πω τελικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στα πλαίσια του θέματος αυτού ε, δεν είναι σκόπιμο να συζητάμε μόνο για τη Δανία. Είναι τα περισσότερα κράτη-μέλη που συνεχίζουν την πρακτική αυτή. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την νομοθεσία και δεν ξέρουν και γιατί πρέπει να το κάνουν, δεν καταλαβαίνουν. είναι σαν ένα ξέφραγο αμπέλι εδώ πέρα αυτή η κατάσταση. Μπαίνει ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Ε, θα πρέπει οι χώρε να συμμορφώνονται με την νομοθεσία και όσοι δεν το πράττουν να υφίστανται τι κυρώσει. Έτσι θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα και θα έχουμε μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει. Είναι θέμα της Επιτροπής Αναφορών αυτό, αλλά παρακαλώ να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση από πλευρά κρατών μελών διότι ο νεοφώτιστος υπουργός κινδυνεύει να ξαναπέσει στον δρόμο της αμαρτίας αν δεν τον βοηθήσουμε να προχωρήσει και να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Όσο Η Πρόεδρος. Θέλω να δώσω το λόγο και στον Πέτερ Γιάρ που το παρακολουθεί αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι είναι παράδειγμα αυτό κακής ευρωπαϊκής Νομοθεσία και θα πρέπει να φροντίσουμε οι ευρωπαϊκοί νόμοι όχι απλώς να αποφασίζονται και να ψηφίζονται αλλά και να εφαρμόζονται. Και με ενοχλεί πάρα πολύ ε, αυτό, γιατί οποίο ξέρει πώς γεννήθηκε αυτό το θέμα, θυμάμαι καλά, είχαμε τριμερή διάλογο και αν θυμάμαι καλά τι είναι τριμερής διάλογος, είναι τρεις. Ε, συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν και νομοθετούν. Δεν, είναι, δεν μπορεί να βγαίνει το κάθε κράτος και να λέει καλά κάποτε κάνω ένα νόμο και σιγά μην τον εφαρμόσω. Και πολύ χειρότερα συμβαίνουν και στη Γερμανία. Λες και οι Βρυξέλλες είναι κανένας μπαμπούλας και μας επιβάλλουν νομοθεσία. Ε, η νόμοι είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού και γι' αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ, με εκνευρίζει πάρα πολύ η κατάσταση αυτή σημαίνει που είναι τόσο στρεβλή. Είναι αυτό. Δεύτερον, έχουμε αφήσει και μεταβατικές περιόδους. Και αν θυμάμαι καλά, δέκα χρόνια. Δηλαδή μετά από 10 χρόνια ε, κάθε εκτροφή έχει αποσβέσει τον εξοπλισμό της, άρα μπορεί να τον ανανεώνει. Ε, και μπορούν να προσαρμοστούν οι εκτροφές και τα χειροστάσια ε, ώστε να μην χρειάζεται να κόβουν τις ουρές των χειριδίων. Για μένα υπάρχουν δύο τινά. Είτε ισχύει ο νόμος και τον εφαρμόζουμε, είτε δεν τον εφαρμόζουμε αλλά πρέπει να αλλάξει. Διότι δεν είναι αποτελεσματικός. Πάντως εγώ πιστεύω ότι είχαμε ε, λόγους αρκετούς και προφανείς να νομοθετήσουμε. Μπορεί η κυρία Άουκεν να ε, εκπλαγεί. Δεν μου αρέσει να κρατάω ανοιχτέ αναφορέ, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω επιβάλλεται. Και μια σύσταση, παράκληση, απέτηση ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Ισχύουν όμω ή δεν ισχύει. Φτάνουν τα λόγια, έργα χρειάζονται τώρα. Τώρα επειδή δεν θέλουμε να πατήσουμε κανένα κάλο, τι θα γίνει, δεν θα προχωρήσουμε για να μην ε, στριμώξουμε κανένα, για να μην πονέσουμε κανένα και πονάμε τους χείρους. Δεν διαμορφώνουμε έτσι, ούτε χτίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε εμπιστοσύνη ανακτούμε. Ε, αγωνιστείτε παρακαλώ από την Κομισιόν και απαιτήστε επιτέλους από τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόσουν. Γιατί δεν μπορεί η εξαίρεση να γίνει κανόνας, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτερ. Και τώρα έχω τον κύριο Κόφου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω δανέζικα ή αγγλικά. Δεν το έχω αποφασίσει. Ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση. Οι συναδελφοί μου το είπαν ήδη. Είναι εσχρό. Απαράδεκτο το να έχουμε αυτή τη στιγμή μια οδηγία που δεν υλοποιείται εδώ και χρόνια από τα κράτη-μέλη. Κοιτάω τώρα, για παράδειγμα, τον τελευταίο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις κάτω από την Επιτροπή, όπου καθίσταται σαφές ε, στα πορίσματα ότι σχεδόν το 100% των χειριδίων ε, στο 100% των χειριδίων ε, κόβουν την ουρά. Και ο λόγος που δεν έχει υλοποιηθεί Ε, αναφέρεται ότι είναι λόγια ανταγωνισμού, όπως είπατε και εσείς. Αν αυτή είναι η δικαιολογία, και όπως είπε και η Μαγκρέτε, ρώτησα και για άλλες χώρες στην Ευρώπη, νομίζω ότι οι περισσότερες χώρες παραβιάζουν την νομοθεσία αυτή. Ε, απαράδεκτο, πραγματικά. Έχω και μια ερώτηση. Αν κοιτάξει κανείς το κείμενο, και αυτό ήταν στην πρώτη ε, κουκίδα της πρώτης διαφάνειας της παρουσίασης, αν δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στη Δανία, εκεί λένε ότι οι γεωργοί πρέπει να προσπαθήσουν να αποφύγουν, να αποτρέψουν το δάγκωμα των ορών. Ε, ναι, αυτοί λένε ότι το έχουν κάνει. Υπάρχει ένα τεράστιο νομικό κενό εδώ, γιατί λένε πάντα, ναι, προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε, οπότε κόβουμε τις ουρές και συνεχίζουμε με αυτή την πρακτική. Οπότε πρέπει να είμαστε σαφείς Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των χείρων και των χειριδίων στην Ευρώπη ή απλά φτιάχνουμε ένα νόμο ο οποίος δεν τηρείται. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Νομίζω ότι η πρόθεση ήταν σαφής. Θέλουμε να ε, ε, προλαμβάνουμε την τακτική ε, τη συνήθη κοπή των ουρών των χειριδίων για να βελτιωθεί η καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά υπάρχουν πολλά παραθυράκια, πολλά κενά και από την Κομισιόν συχνά ακούμε, ναι, ξέρετε, υπάρχουν παραθυράκια, ναι, δεν έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση νομοθεσία. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα ήθελα να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή. Ναι, φαντάζομαι αν αυτό ήταν ο τομέα των χρηματοοικονομικών. Φανταστείτε. Αν τώρα μιλάμε για τον τραπεζικό τομέα, για κάτι που σχετίζεται με τα χρηματοοικονομικά, θα είχαν ακολουθήσει διαδικασίες σε παραβάση τάχιστα. Ενώ εδώ μιλάμε για ζωντανά όντα, για χειρίδια, για μικρά γουρνάκια τα οποία συστηματικά τους κόβουν τις ουρές τους και τα μεταχειρίζονται με έναν απαράδεκτο τρόπο. Για μένα αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ε, απαράδεκτης κατάστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αποτρόπαιο το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν θέλει... Εντάξει, να έχετε κάνει πολλά πράγματα, αλλά το πράγμα μιλάει από μόνο του. Εδώ μιλάμε τη γλώσσα του χρήματος ουσιαστικά. Ε, διαδικασίες σε παραβάση, θα κόστιζαν πολύ για τα κράτη-μέλη ε, και θα είχαν βέβαια και αποτέλεσμα. Τέλο πάντων, να δώσω ξανά το λόγο στου ε, αναφορείς πολύ σύντομα για να μας πείτε τη σκέψη σας, τι θα θέλετε να κάνουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε και προφανώς υπάρχει συνένεση στο στα μέλη της Επιτροπής σας για να μείνει η αναφορά αυτή ανοιχτή και έχετε απόλυτο δίκιο. Όντως εδώ είμαστε η ντροπή της Ευρώπης γιατί νομίζω ότι πρόκειται για ε, προσπάθεια κοροϊδίας της εξαιρετικής νομοθεσίας για την ζωή των ζώων την οποία εμείς δεν τηρούμε. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία να τη βελτιώσουμε. Επίσης, Πολύ συχνά λέμε πως έχουμε τα ισχυρότερα πρότυπα για την ε, ζωή των ζώων σε όλο τον πλανήτη. Όμως όταν ε, διαπραγματευόμαστε εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους μας βλέπουμε ότι και ήδη ξέρουν πως οι ίδιοι τους κανόνες που προσπαθούμε να προωθήσουμε δεν τους στηρούμε. Άρα γιατί να μας αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα. Και αν πραγματικά δεν μπορούμε αυτή την νομοθεσία να την εφαρμόσουμε, γιατί τι είδους ισχυρά πρότυπα ε, μιλάμε. Χαίρομαι γιατί η δική σας ισχυρή θέση θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να πιέσει τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Φρέντρικ. Ε, ευχαριστώ και θα συμφωνήσω απόλυτα. Τουλάχιστον όλα τα μέλη που είμαστε εδώ νομίζω ε, αντιμετωπίζουμε μεγάλη συνένεση το θέμα αυτό, ομόφωνα θα έλεγα και θα το ξεκαθαρίσω. Πιστεύω πως ο Επίτροπος κ. Ανδρουκάητης έχει κάθε καλή πρόθεση. Όμως, επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προτείνει περισσότερη νομοθεσία από ό,τι χρειάζεται, δεν καταφέρνει να φέρει σε πέρα σε αυτό που επιθυμεί, γιατί ξέρετε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρέχουσα στρατηγική για την ε, ευζοία των ζώων αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αυτά τα οποία νομοθετήθηκαν πριν από μερικά χρόνια και αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε τις τελευταίες νομοθετικές ε, διατάξεις. Τίποτα δεν βρίσκεται στα σκαριά και λυπάμαι πολύ που θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι γιατί ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος οποίο δεν θέλει να δράσει, αλλά γιατί είναι συλλογικό όργανο το Κολέγιο των Επιτρόπων και πρέπει να το αποφασίσουν από κοινού. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλη τη συνέβη πριν από δύο χρόνια με το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήταν ένα αρκετά απλό ψήφισμα που ζήτησε όμως μια νέα στρατηγική για το θέμα αυτό για τα επόμενα 4-5 χρόνια και θέλαμε συμμόρφωση με τους κανόνες που έχουν ήδη θεσπιστεί Και τελικά, νομίζω πως φτάσαμε στην κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε για μια νομοθεσία για την προστασία των ζώων που ε, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο τα νοήμωνα ζώα. Ε, και νομίζω έχουμε και την έκθεση Πόλσεν, η οποία για πρώτη φορά στην παγκόσμια νομοθεσία η Ευρώπη ανέλαβε ε, τον ηγητικό ρόλο και είπε πως είναι νοήμωνα όντα τα ζώα. Και αυτός είναι ένας τρόπος που μας επιτρέπει την νομοθετική μας εργασία να την προωθήσουμε προς μια άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή αν θεωρούμε πως δεν είναι νοήμονα ζώα, πως αν δεν αισθάνονται ε, τα ζώα ε, τον πόνο, τότε θα είναι τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Μάργαρετ, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δω τον κατάλογο αυτών των χωρών γιατί πάντα λέμε οι περισσότερε χώρε και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν χώρε οι οποίε συμμορφώνονται με του κανόνε. Και θα ήθελα να δω ποιε είναι. και να σας πω πως είναι πραγματικά καταθλιπτικό σε κάποιο βαθμό γιατί το Arhaus, το Πανεπιστήμιο του Άρχαους παρουσίασε μία μελέτη που λέει 100 κιλά χείρος 1,2 τετραγωνικά μέτρα ε, χώρος και 150 γραμμάρια σανό κάθε μέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά υποχρεωτική κοπή. Γιατί αν δείτε τους χείρους πώς ζουν και πώς ζουν όταν είναι ελεύθεροι, είναι καταπληκτικοί. Ζούνε και παίζουν και σε πειράματα που έχουν γίνει, γιατί έγινε μια σχετική εκθέση, χρειάζονται κάθε τρίτη μέρα καινούριο, ε, καινούργια παιχνίδια ε, και πρέπει να σου πω πω κάθε, κάθε τρεις είχαν εξαντλήσει τη δυνατότητα κάθε παιχνιδιού που του δίναμε και περιμέναμε να του φέρουμε κάτι καινούριο. Οπότε καταλαβαίνετε το 1,2 τετραγωνικά μέτρα και τα 150 γραμμάρια σαν την ημέρα δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ναι, όταν υπάρχει πρόθεση υπάρχει και τρόπος. Κύριε Τζίλ. Ευχαριστώ πολύ. Στη βορειοανατολική Αγγλία όπου η χειροτροφία είναι εντατική. Γνωρίζω πολλούς γεωργούς οι οποίοι χρεοκόπησαν διότι όταν τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για την ε, καλή μεταχείριση των ζώων συμμορφώθηκαν ενώ οι άλλοι αγρότες στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν το έπραξαν και έτσι ε, απαιτήθηκε να ανταγωνιστούν με αθέμητο τρόπο και αυτό που αφορά ε, τους Βρετανούς ε, σε σχέση με την Ευρώπη είναι ότι υπέθεταν ότι η Ευρώπη είχε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού αυτό δεν συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο πολλοί αγρότες ψήφισαν υπέρ του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι αντιλήφθηκαν ότι ήταν άδικος ο τρόπος που λειτουργούσε. Ένας τρόπος που μπορούμε να βελτιώσουμε τη μεταχείριση των ζώων είναι ένα συνεκτικό σύστημα επισήμανσης ώστε οι καταναλωτές να αποφασίζουν αυτοί με τις τσέπες τους αν επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα τα οποία έχουν εκτραφεί σε ένα περιβάλλον καλής μεταχείρισης ε, και σε ένα περιβάλλον όπου η σφαγή έχει γίνει με ένα σωστό τρόπο. Διότι πολλοί κόσμος πάει και τρώει ε, μπέργκερ από τα McDonald's χωρίς να καταλαβαίνουν ότι τα ζώα αυτά έχουν σφαγεί με τρόπους ε, απαράδεκτους ή ότι έχουν σφαγεί με τρόπο χαλάλ. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μεταχείριση των ζώων δίνοντας την επιλογή αυτή στον καταναλωτή, ο οποίος πιστεύω ο Ευρωπαϊο καταναλωτός θα πληρώσει λίγο παραπάνω, θα αγοράσει με την καρδιά του ώστε να είναι βέβαιος ότι έχουν χρησιμοποιηθεί διαδικασίες καλύτερης μεταχείρισης των ζώων στο κρέα που τρώει. Οπότε ας δούμε αν μπορούμε να βάλουμε μια ετικέτα, μια επισήμανση, ώστε να υπάρχουν ισές συνθήκε ανταγωνισμού. Πρόεδρο, ωραία. Α μην το συνεχίσουμε τώρα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε ω πρόταση, να την εξετάσουμε. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Φυσικά θα διατηρήσουμε τι αναφορέ ανοιχτέ. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα έχουμε επιχείρηση να στείλουμε μια επιστολή στον Επίτροπο Αντριουκάητη. Ελήφθη, ε, μα έχει απαντήσει και πιστεύω ότι πρέπει να την ξαναστείλουμε αναφέροντα την τρέχουσα κατάσταση όπω έχει σήμερα. Δεν θέλουμε παραπάνω νομοθεσία, απλά θέλουμε η υπάρχουσα νομοθεσία, η υπάρχουσα οδηγία να υλοποιηθεί παντού. Και η Κομισιόν να παρακολουθεί την υλοποίηση. Καλό θα ήταν λοιπόν να κατανομάσουμε τις χώρες αυτές που δεν ε, ε, υλοποιούν σωστά, δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία. Πέραν αυτού θα ήθελα να σας ζητήσω να κάνουμε και κάτι που δεν κάνουμε συχνά. Να στείλουμε μια επιστολή στην Προεδρία του Συμβουλίου. Οι Βούλγαροι αυτή τη στιγμή κατέχουν την Προεδρία του Συμβουλίου και θα μας ενδιαφέρει να δούμε την αντίδρασή τους. αν τη στείλουμε, θα χρειαστεί να το συζητήσουν υποχρεωτικά με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια καλή ιδέα και βλέπω ότι μου γνέφουν οι συνάδελφοι. Μερικέ φορέ καλό είναι να είμαστε λίγο δημιουργικοί, αν και πολιτικοί ε, όπως κάναμε και σήμερα. Ωραία λοιπόν. Ε, και για να επανέλθω τώρα σε αυτό που είπε η Μάργκρετ για τα σχήρους, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ζώο τόσο κοντινό στον άνθρωπο όσο τα γουρούνια, όσο οι χείροι. Και εμεί μερικέ φορέ βαριόμαστε, αλλά σήμερα σε αυτή την επιτροπή δεν βαριόμαστε. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτέ είναι πολύ σημαντικέ αναφορέ και τώρα έχουμε μια οδό που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ όλου σα. Βλέπω ότι μου γνέφετε όλοι. Οπότε ολοκληρώνουμε με, αυτό το θετικό, ε, με αυτή τη θετική νότα, με αυτό το θετικό πνεύμα. Και ευχαριστώ και τους αναφέροντες που μας διαφώτισαν. Ευχαριστούμε πολύ. It's not possible. Okay. So we move to the next petition which is 1212. Να περάσουμε λοιπόν στη 1212 που είναι τα προβλήματα που είχαν τα βοηδή με τα ενότια ταυτοποίηση στην Ιρλανδία. Νομίζω ότι έχουμε εδώ μια ομάδα αναφερόμενων από την Ιρλανδία. Πάντως οι αναφέροντες οι οποίοι υπέβαλαν αυτή την αναφορά δεν ε, είναι στην αίθουσα, οπότε να δώσω το λόγο απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Κέλλη, εσείς εκπροσωπείτε τους αναφέροντες. Δεν το ήξερα. Ε, σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και είμαι εδώ με τον Τόμ και τα παιδιά του, τον Τζον και την Πατρίσια, οι οποίοι υποβάλλουν αυτή την υπόθεση και ήθελα να σας πω πως εγώ θαυμάζω ιδιαίτερα την Επιτροπή Αναφορών, κάνουν πολύ καλή δουλειά και δεν φέρνω εγώ εδώ αναφορές έτσι εύκολα και ήταν η πρώτη φορά που το έκανα ε, τέσσερα χρόνια πριν όπου είχαμε ένα ε, σημείο με τοξικά απόβλητα στην περιοχή του Κόρκ με μεγάλο, που είχε τεράστιες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και πρέπει να σας πω ότι μετά την αναφορά αυτή η κυβέρνηση έκανε ό,τι έπρεπε, αποκαταστάθηκε η περιοχή και πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Σήμερα είναι εξίσου σημαντικό το θέμα ε, και κυρίως για τους ε, ε, αναφέροντες και ο Τόμ που είναι εδώ και έχει να κάνει με το σύστημα ταυτοποίησης βοηδών. Δηλαδή με τα ενότια που φορούν. Ο Τόμ και η γυναίκα του ημέρη είχαν δύο διαφορετικές εκμεταλλεύσεις, δύο διαφορετικά κοπάδια με διαφορετικό αναγνωριστικό αριθμό. Κανένα πρόβλημα. Και ένας πολύ γνωστός συγγραφέας διηγημάτων, ο Κόνορ, στην Ιρλανδία είπε πως τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα. Και να σας πω πότε ξεκίνησαν εδώ όλα τα προβλήματα. Όταν, όταν πέθανε η πεθερά του Τόμ, καθάρισαν το σπίτι και 30 ενότια τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί πετάχθηκαν και καταστράφηκαν. Δεν έδωσαν σημασία και στο συνεταιρισμό ε, στην περιοχή τους ζήτησαν να τους δώσουν καινούργια νότια την επόμενη χρονιά. Τελικά όμως τους είπαν το Υπουργείο Γεωργίας ε, τους είχε πει στο συνεταιρισμό να μην τους δώσουν επιπλέον ενότια γιατί τους περίσβαν ενότια από προηγούμενες χρονιές και δεν θα μπορούσαν να τις, ε, και δεν χρειαζόντουσαν επιπλέον. Οπότε δεν τους δώσανε ενότια εκείνη τη χρονιά, είχαν ε, γεννήσεις βοηδών, δεν μπόρεσαν να τα καταχωρήσουν στο Μητρό όπως πρέπει και ήρθαν σε επαφή με το Υπουργείο Γεωργίας και καμιά φορά τους τηλεφωνούσαν τρεις ε, μέρες και ήταν ε, την εποχή που ξέσπασε ο αυθόδης πυρετός στην Ιρλανδία. Ήταν μια δύσκολη εποχή. Και ίσως το Υπουργείο, τι να σας πω, στάθηκε ιδιαίτερα προσεκτικό, προσπάθησε να εφαρμόσει με υπερβολική αυστηρότητα τους κανόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν υπερβολικά προσεκτική και πρέπει να πω ότι μάλλον ε, άκομψα φέρθηκαν στον Τόμ και τη Μέρη με αποτέλεσμα να έχουν βοηθεί στην εκμετάλλευση χωρίς να έχουν ενότια να τους φορέσουν, χωρίς να μπορούν να τα καταχωρήσουν, χωρίς να μπορούν να τα πουλήσουν. Και έφτασε ο χειμώνα και δεν είχαν και αρκετά, αρκετές, αρκετά, αρκετή ζωοτροφή για να τα ταΐσουν. Οπότε Συνεχίστηκε έτσι η κατάσταση χωρίς να δοθεί μια λύση και τελικά το Υπουργείο είπε ότι εντάξει θα κάνει τεστ DNA ε, στα ε, καινούργια βοηθή που είχαν γεννηθεί έτσι ώστε να φανεί ποια είναι η μητέρα τους και αυτό ήταν εύκολο γιατί είχαν πια μεγαλώσει Αλλά βέβαια η οικογένεια υπέφερε γιατί για παράδειγμα ήρθε κάποιος υπάλληλος του Υπουργείου και του είπε ότι εγώ ε, θα τα θανατώσω τα ζώα γιατί δεν ε, έχουν τα κτλ. Και ήταν μια φρικτή κατάσταση και τελικά η Ένωση Κτηνοτρόφων της Ιρλανδίας δεν ε, ε, ε άντεξε έχασαν την πρώτη δίκη, πήγαν στο διαμεσολαβητή, ήρθαν σε μένα, του είπαν ναι, είναι όντω άδικο και ελπίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών θα υποβάλει μια σύσταση έτσι ώστε τέτοιε περιπτώσει να τι μεταχειρίζονται με άλλο τρόπο. Τώρα το κομβικό σημείο εδώ είναι το εξή. ότι δυστυχώ συμβαίνουν συμπτώσει στη ζωή. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Τα τρία χρόνια που συνεχίστηκε αυτή η υπόθεση 2000, 2001 και 2002 ήταν οι χρονιές αναφοράς για να δοθούν τα δικαιώματα στα διάφορα καθεστώτα και για να πληρωθούν οι πρημοδοτήσεις. Οπότε το γεγονός πως δεν μπορούσε να κατοχωρήσει τα βοηθή του οτόμ εκείνης τι της χρονιές οδήγησε τον, ε, την άνοιξη του 2003 να μην μπορεί να αιτηθεί γιατί δεν μπορούσε να καταχωρήσει τα βοηθή, δεν μπορούσε να πληρωθεί τις πρημοδοτήσεις και έκτοτε κάθε χρόνο έχει οικονομική απώλεια η οποία σωρευτικά φτάνει στον ένα τεράστιο ποσό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν έλαβε αυτές τις πρημοδοτήσεις τον οδήγησε ε, στο να κλείσει ένα κομμάτι της ε, ε, εκμετάλλευσης, έβαλε υποθήκη, έχει πρόβλημα με την τράπεζα. Οπότε οι μέρη και αυτός υπέφεραν πάρα πολύ ως αποτέλεσμα αυτής της τακτικής. Και νομίζω πως το Υπουργείο ΜΕΝ ήταν υπερβολικά αυστηρό για να εξασφαλίσει πως όλοι θα συμμορφωθούν με το γράμμα του νόμου, γιατί ναι, στην Ευρώπη και στην Ιρλανδία λέμε πως έχουμε ιχνηλασιμότητα. Ναι, από, το, ε, από την εκμετάλλευση μέχρι το πιάτο. Αλλά εδώ, δεν, ε, εδώ χάθηκε η κοινή λογική. Και εντάξει, έγινε μια πραγματική προσπάθεια. Έγινε ένα ατυχές λάθος. Πετάχτηκαν τα ενότια. Μα δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Δεν φάνηκε κάπου να υπάρχει κάποιο ζώο με το ενότιο αυτό. Όλα τα ζώα βρέθηκαν στην εκμετάλλευση όταν δόθηκε μια λύση και τελικά κάπως λύθηκε. Οπότε δεν υπήρχε ούτε καν υπόνοια απάτης, δεν προσπάθησαν ε, κάποιον να κοροϊδέψουν. Ήταν μια τυχής σύμπτωση η οποία δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Και ο Τόμ και η Μέρη υπέφεραν πάρα πολύ ως αποτέλεσμα αυτής. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ λογικό και πολύ δίκαιο να λέμε πως είχαν δικαίωμα να λάβουν αυτές τις πληρωμές για τις περιόδους αναφοράς και θα έπρεπε αυτά τα χρήματα, αυτές οι ενισχύσεις να τους καταβληθούν τώρα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο. Και δεν βλέπω να υπάρχει οποιαδήποτε λογική στο να μην τους πληρώνονται αυτές οι ενισχύσεις γιατί τα βοηθοί υπήρχαν. Ναι, τελικά καταχωρήθηκαν και επειδή απλώς δεν ήταν καταχωρημένα τη στιγμή της περίοδου αναφοράς, χάθηκαν πρημοδοτήσει. και πρέπει να σας πω ότι με όλα αυτά δεν μπορούσαν καν να αγοράσουν και καινούργια ζώα οπότε είχαν μπει σε έναν αδυσόπιτο κύκλο νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτό και αν έχετε ερωτήσεις με χαρά θα απαντήσουμε yeah, να συμπληρώσει τίποτα ε, πραγματικά όλα αυτά συνέβησαν το 2000, ε, μάλλον 26 αγελάδες είχα ε, και 85 ε, δικαιώμουν σε τρία χρόνια να σε αυτά. Και εκτός αυτού αφαίρεσαν και την άδεια που έχει η γυναίκα μου που ήταν 300 χρόνια αγρότες η οικογένειά της και δεν έχει κάνει ε, κανένα έγκλημα ούτε δόλο είχε ούτε τίποτα και της αφαίρεσαν τον αριθμό αδειοδότησης μετά από τόσες γενιές ε, εκμετάλλευσης και ε, αγροτίας. Είναι πραγματικά ε, τρομερά αυτά που κάνουν στο Υπουργείο Γεωργίας. Και αρκετά, κάτι άλλο κύριο Σκέλη. Ο Τόμι είναι διάσημος πια στην Ιρλανδία γιατί η ίδια η Ελλάδα του πέρυσι γέννησε τέσσερα μοσχάρια τετράδημα. Ναι. Και βγήκε και στην τηλεόραση τον Αύγουστο και στις ειδήσει και δεν έχει πάρει ακόμα τα λεφτά που του χρωστάνε. Αλλά τι να την κάνει τη διασημότητα αν είσαι φτωχό, ε, βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον, συγχαρητήρια για τα τετράδημα. Ελπίζω κάποια στιγμή να ανταμυφθείτε γι' αυτό. Λοιπόν, ε, θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μποζού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι γεγονός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε αυτή την αναφορά και επιβεβαιώνει ότι η κατάσταση ε, όπως περιγράφει ε, είναι ε, ακριβής. Όταν συνέβησαν αυτά υπήρχε ε, υποχρέωση ταυτοποίηση και αναγνώριση των βοηδών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτά είναι στη Γενική Διεύθυνση ε, ε, δημόσια και προστασία του καταναλωτή για να μπορείς να αναβάνεις τις που είναι κατά κεφαλή ζώου στην εκτροφή, για τη βοτροφία και ανάλογα με την νομοθεσία και σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Είναι γεγονός ότι ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν τα ζώα δεν ήταν επιλέξιμη εκτροφή για τις πρημοδοτήσεις και τα δικαιώματα σπληρωμές μετά από την ε, αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2003 όπου αποσυνδέθηκαν μεν οι ενισχύσεις από την παραγωγή αλλά για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς ε, λαμβανόντουσαν υπόψη για τον υπολογισμό των ποσών. Και βεβαίως αν δεν ήταν τα ζώα επιλέξιμα αυτό επηρέασε και τα δικαιώματα και τον υπολογισμό τους. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να θυμίσει ότι εδώ πρόκειται για ε, συνυπευθυνότητα, δηλαδή τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα και την εξουσία να ελέγχουν την κάθε περίπτωση και να εκχωρούν τα δικαιώματα. Η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ε, να έχει σχέση με ένα διοικητικό πρόβλημα και όχι με τρόπο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θλίβεται μεν για την κατάσταση αυτή, πλην όμως έχει περιορισμένες δυνατότητες δράσης και θα θέλαμε να συστήσουμε στους αναφέροντες να αποταθούν στην εθνική δικαιοσύνη αν έχετε εξαντλήσει όλες τις διοικητικές οδούς Βεβαίω, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αυτό το θέμα. Δεν μπορώ δυστυχώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ε, συνάδελφοι, ο Πέτα για... Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα διαπιστώσατε ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο όταν είσαι βόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το να μην έχει ενότιο. Έχουμε πάρα πολύ ε, περιοριστικό σύστημα ταυτοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το είδαμε και στο προηγουμένο, ε, προηγούμενο θέμα με τα χειρίδια, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που κάνουν τα κράτη-μέλη ό,τι τους καπνίσει και τώρα έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. 100% ε, πρέπει να τηρηθεί η νομοθεσία με τρόπο σχολαστικό στη βοοτροφία. Και άλλο παράδειγμα έχουμε έχουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου του ευρωπαϊκού στις άμεσες πληρωμές είναι κάτω από 2% το ποσοστό σφάλματος και θαυμάσια είναι όλα αυτά και πολύ ωραία. Δηλαδή είμαστε κάτω από το στατιστικό λάθος. Σχεδόν κανένα σφάλμα δεν έχουμε. Το πρόβλημα ποιο είναι στο σύστημα. Και ε, γιατί θέλω να το ερμηνεύσω, γιατί αναρωτιέται κανείς πώς γίνεται αυτά τα πράγματα, γιατί το κάνουν οι τοπικές αρχές. Γιατί το κάνουν... Ε, αυτό σε έναν ε, εκτροφέα και ο άνθρωπος δεν τα έχει εφεύρει ε, τα βοηδή υπάρχουν εκεί, μπορείς να τις πιάσεις γελάδες έχουν χάσει την ταυτότητά τους, έχουν χάσει το ενότιο αυτό το σκουλαρίκι που φοράνε και υπάρχει ένα συστημικό λάθος που έρχεται να προσθεθεί ότι είναι τόσο στενός κορσές το σύστημα. Αν κάνει κάποιο λάθος μια τοπική αρχή και το διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, θα πρέπει να επιστρέψει τα κονδύλια που πήρε ως μειόφιλη η χώρα ε, αχρεωστήτως καταβληθέντα αλλά τους το καταλογίζουν και ως απάτη. Οπότε φοβούνται και τη σκιά τους οι τοπικές αρχές. Ε, δηλαδή να μην κάνουν τίποτα μετά την υποδιαστολή γιατί σε περίπτωση που γίνει το παραμικρό θα βρούνε τον πελά Γιατί μπορεί ο αγρότης να χρειαστεί να επιστρέψει 10.000 και το κράτος 20 εκατομμύρια και θα έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό είμαστε στο σφάλμα στο 2% γιατί φοβούνται και τη σκιά τους και δεν κουνιούνται καν. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από ό,τι φαίνεται επί τόπου να ρυθμιστούν προβλήματα μιας μεμονωμένη αγέλη. Γιατί σου λέει άλλος καλά δεν μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα και η κυκλοφορία αφορά τόσα χρόνια. Κανονικά από τις Βρυξέλλες λένε ότι πήγαν όλα καλά και να το αριθμίσουν οι τοπικές αρχές. Οι τοπικές αρχές τρέμουν ε, και είναι σε φαύλο κύκλο ο αγρότη. Τώρα, ε, να στείλουμε γράμμα στον Επίτροπο, γενικά στι άμεσε πληρωμέ έχω πρόβλημα το ξέρω ότι δεν σας παρηγορεί αυτό που λέω. Δεν είστε μόνο σας στην Ευρώπη όμως ε, που έχετε τέτοιες συμφορές χωρίς κακή πρόθεση και χωρίς να έχετε κάνει τίποτα κακό βρίσκεται απέναντι την νομοθεσία και έτσι αποφασίζουν τα Υπουργεία και οι αρχές. Θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση για τέτοιες περιπτώσεις που να μπορεί κάποιος να αποφασίσει. Ενία δεν υπάρχει αυτό. Άλλο έναν αριθμό να σας δώσω. Λένε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Ναι, αλλά 40 δισεκατομμύρια είναι άμεσες πληρωμές προς τους αγρότες. 1,5% για δεν ξέρω ποιο λόγο δεν απορροφώνται. Δεν είναι καν οικονομικό το πρόβλημα. Το προηγούμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είπαμε πώς είναι δυνατόν κάνουμε νομοθεσίες και τις αψηφούν όλοι. Τώρα είναι το ανάποδο. Έχουμε κάνει τόσο περιοριστικό αυτό το πλαίσιο που δεν έχει κανένα περιθώριο λιγμών κάποιος που θέλει να διορθώσει μια στρεβλή κατάσταση. θα πρέπει να υπάρξει μια επιτροπή σοφών, δεν ξέρω μυτική πώς να λέγεται, που να ρυθμίζει αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις όταν κάτι πάει στραβά. Από τη σκοπιά των Βρυξελών είναι όλα αυτά μακριά και όποιο είναι έξω από το χώρο πολλά τραγούδια ξέρει. Ε, γιατί σου λέει τώρα πενταροδακάρι. Ναι, για τι Βρυξέλλε μπορεί να είναι λίγα τα λεφτά, για τον άνθρωπο μπορεί να είναι καταστροφή του. Γιατί δεν υπάρχει μια ρύθμιση για έκτακτε περιπτώσει, όταν κάτι πάει στραβά για τον οποιοδήποτε λόγο να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έχει πληγεί και να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για το σύστημά μας, για το περιθώριο σφάλματος, αλλά καθόλου περήφανοι για το πώς ε, λύνουμε κάποια λάθη που έγιναν για λόγους αβεβαιότητας, για λόγους αντικσοότητας. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός. Και τελικά πού οδηγεί αυτό. Έχουμε μια επιτυχή κοινή γεωργική πολιτική, αλλά αυτά τα παραδείγματα μας καταστρέφουν αυτή την επιτυχία, γιατί βγαίνει ο ενδιαφερόμενος ή ο πληγής και σου λέει «Μα τι κάνουν αυτές τις Βρυξέλλες, ρε παιδάκι μου». Και δεν αφορά μόνο εσάς αυτό, αλλά και άλλες ιστορίες που είναι σε διέξοδο. Κύριε Τζίλ. Ναι, ευχαριστώ, Τόμ. Αντιλαμβάνομαι την κατάστασή σας και συμπάσχω. Πιστεύω ότι δεν είστε όμως μόνος. Το ζήτημα αυτό ε, εμφανιστήκε και στην Οαλία όταν βγήκε η ID ε, Ανησύχησε όλους τους αγρότες, διότι αν το σκεφτείτε η μέση ηλικία ενός αγρότη ήταν πάνω από 70 και όχι μόνο είχαν να τρέξουν τι επιχειρήσει του, να ασχοληθούν με όλα τα χημικά και τι νέε νομοθεσίε και όλα αυτά, αλλά έπρεπε να βρουν τώρα πλέον και ένα νέο τρόπο σήμανση ε, των ζώων, χείρων, ε, αγελάδων που καμιά φορά έβγαζαν μόνα του τι επισημάνσει αυτέ και καταστρέφονταν. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουν υπολογιστέ που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του. Το ζήτημα είναι ότι πολύ γρήγορα η ζωή έγινε πάρα πολύ δύσκολη για πάρα πολλούς αγρότες ε, που είναι αυτόνομες οντότητες ουσιαστικά και όπως με όλες τις νομοθεσίες υπήρξαν ανεπιθύμητες ε, συνέπειες όπως συνέβη στον ΤΟΜ. Κανείς δεν σκέφτηκε διεξοδικά όλες τις συνέπειες. Κανεί δεν σκέφτηκε να επιτρέψει στα Υπουργεία ε, να προσδώσει κάποια ευελιξία στα Υπουργεία Γεωργία των διαφορών χώρων. Πρέπει να υπάρχει μια κοινή λογική και το πρόβλημα είναι ότι η κοινή λογική δεν απαντάται κοινά. Δεν απαντάται συνήθω. Ε, όταν φοβάται το Υπουργείο να λάβει μια απόφαση, ε, μήπω και χάσει τη δουλειά του ο συγκεκριμένος υπάλληλο Τι πρέπει να γίνει, πρέπει να μιλήσουμε στην Επιτροπή Άγκρη, σε ποια Επιτροπή, σε ποιον πρέπει να μιλήσουμε ώστε να μην επαναληφθεί αυτό. Κατά την άποψή μου πρέπει ομόφωνα όλοι να δείξουμε μεγαλοψυχία ε, προς τον Τόμα και προς ε, όλους τους άλλους ανθρώπους που κάνουν μια τόσο δύσκολη δουλειά και να του πούμε ναι, είμαστε οι μεγάλοι, αλλά θα μείνουμε στο πλευρό των μικρών και θα φροντίσουμε να λάβετε αποζημίωση αυτό που σας αξίζει. Το ξέρω αυτό από ιδέα εμπειρία. Έχω μιλήσει με πολλούς αγρότες που είχαν προβλήματα με, αυτές τις, ε, με αυτά τα ενότια. Είναι εφιάλτης και είναι το τελευταίο που θέλει κανείς όταν βρίσκεται στο χείλο του γκρεμού, στο χείλο της χρεοκοπίας να... Ε, για να βρει κάτι που να αξίζει περισσότερο από την ε, δουλειά του και ξαφνικά έρχεται κάποιος και απειλεί να πυροβολήσει τα ζώα σας. Είναι απαράδεκτο, ντροπή. Αν είναι να κάνετε ένα πράγμα εδώ, ε, είναι ότι πρέπει να ε, σταθείτε στο πλευρό των πολιτών σας. Δεν, δεν, δεν αναφέρομαι σε εσά προσωπικά ω μικρό άνθρωπο. Δεν είστε μικρό άνθρωπο, φυσικά. Δεν είστε Είστε ένας αγρότης και αυτό είναι ε, φιλοφρόνηση όταν σας το λέω. Είναι... Ο νόμος σε αυτή την περίπτωση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Θέλαμε να υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση και ακούμε ε, συνεχώς πολιτικούς να μιλάνε για δικαιοσύνη και εδώ δεν βλέπουμε καμία δικαιοσύνη. Σας έχουν αντιμετωπίσει άδικα και αν έχει οποιαδήποτε εξουσία αυτή εδώ η Επιτροπή να μιλήσει με το Υπουργείο Γεωργίας ε, της Ιρλανδία και να βρει ποιος ασχολήθηκε με αυτή την περίπτωση. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να ε, κάνουμε επίση, επιτέλους κάτι με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πια ότι πρέπει να το αφήσουμε εδώ, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Το Υπουργείο από τις αρχές Μαΐου του 2001 γνώριζε πως ε, τα ζώα είναι στη θέση τους χωρίς να έχουν καταχωρηθεί και χωρίς να έχουν καταγραφεί και χωρίς να φέρουν ενότιο. Αλλά εκείνη τη στιγμή έτρεχε ο αυθόδης και κάθε κάθε γεωργός και κτηνοτρόφος στην Ιρλανδία, επειδή είχε αυθόδη στην ε, ε, Αγγλία, έκανε ό,τι μπορούσε για να ε, προλάβει τον εξαπλωθεί και σε η ασθένεια. Οπότε, εάν υπήρχε οποιοδήποτε μη καταγεγραμμένο ζώο και έπεφτε σε λάθος χέρια, θα μπορούσαμε να έχουμε καταστρέψει την κτηνοτροφία στην Ιρλανδία. Καταλαβαίνετε το βάρος. Και επίσης, έχουμε και μια ενδοϊπηρεσιακή επιστολή όπου λένε πως κάνουν λάθος στο Υπουργείο. και η συγκεκριμένη διατύπωση έλεγε θα έπρεπε να έχουμε ε, δράση νωρίτερα και αν αποτύχουμε θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι και προτείνουμε ότι το Υπουργείο θα πληρώσει για το τεστ DNA και καταλάβετε ότι το Υπουργείο να αναλαμβάνει να πληρώσει ε, δεν θα το έκανε παρά μόνο αν ήξερε ότι είναι υπεύθυνο. Οπότε, αν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, ε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Τζον για τη βοήθεια που με έχει προσφέρει. Σας ευχαριστώ πολύ ε, και σας διαβεβαιώ πως θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας βοηθήσουμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση αυτή και πρέπει να σας πω ότι εγώ θυμάμαι με μεγάλη χαρά τον Ιρλανδό που είχε έρθει στην δική μας επιτροπή απελπισμένος λέγοντας πως δεν θα κάνουμε τίποτα και μετά μου στείλε μια επιστολή και μου είπε νόμιζα ότι θα πάω σε αυτό το μεγάλο κτίριο στις Βρυξέλλες και τελικά με τόση θέρμη με υποδέχτηκαν και ήταν ε, νομίζω ε, δασολόγος ε, κάπου στην ε, επαρχία της Ιρλανδίας και κατάφερε στη μεταγραφή της οδηγίας να κάνει μια διαφορά πώς ως μεμονωμένος πολίτης. Οπότε η Επιτροπή Αναφορών έχει πετύχει πολλά στην Ιρλανδία για τους καθημερινούς ανθρώπους και ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής είμαι εξαιρετικά υπερήφανη και ικανοποιημένη. Και το λέω αυτό για να καταγραφεί στα πρακτικά. Έχουμε κάνει πολλά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Τώρα, να το να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Α, Πίτερ, θέλεις και εσύ να πεις κάτι. Ναι, ήθελα να συμπληρώσω κάτι που είπε ο συνάδελφο. Η Επιτροπή Γεωργίας ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και είναι σύμμαχό μα και στο πλευρό μα. Εγώ θα μιλούσα για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Δηλαδή, είτε ε, θα γίνει μια ε, δικαστική ε, διαδικασία επιτόπου, Αλλιώς δεν μπορούν να τους δώσουν τα χρήματα γιατί είναι ε, παράνομη ενίσχυση. Και είναι σε φαύλο κύκλο εκτεθειμένος μετά ο ε, κτηνοτρόφος. Αυτό είναι το σχισοφρενέζα. Αυτά τα στείλουμε εμείς λοιπόν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, όχι στη Γεωργίας. Γι' αυτό είπαμε, ο στενός κορσές αυτός βοηθάει να είναι κάτω του 2% το σφάλμα και πραγματικά και μπράβο του αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο ε, για να λυθούν πράγματα που πήγανε στραβά. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Τέτοια πράγματα θέλει η Επιτροπή Ελέγχου. Εμείς κάνουμε πολιτική για τους πολίτες, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους και όχι εναντίον τους. Δεν θεωρούμε ότι ο αγρότης μας εξαπατά για να πάρει ενισχύσεις. Ίσα ίσα τον επιβραβεύουμε για αυτό που κάνει για την κοινωνία θα πρέπει να το κοιτάξει η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Υπάρχουν και άλλε μεμονωμένε περιπτώσει που είναι αντίστοιχε για να ξεφύγουν, να σπάσει αυτό ο φαύλο κύκλο. What, Ό,τι μπορούμε ε, να κάνουμε θα το κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει του Κοινοβουλίου, ή μάλλον τον κανονισμό γενικά την νομοθεσία, στην ε, συνυπευθυνότητα ε, τα θέματα των γεωργικών προϋπολογισμών και όλες τις λεπτομέρειες τα χειρίζονται τα κράτη-μέλη. Εκτιμούν την κατάσταση και την περίπτωση και παίρνουν την απόφασή τους ε, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και για τα συστήματα αποζημίωσης. Ακριβώς ε, είναι ένα θέμα κακοδιαχείρισης και κακοδιοίκησης στην Ιρλανδία και μην κατηγορείτε ποτέ ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Να κατηγορήσετε τη χώρα σας και μπορώ να σας βοηθήσω να αποστείλω και άλλη επιστολή, μπορώ να το κάνω. Και επίση η Επιτροπή Γεωργίας έχει ασχοληθεί με αντίστοιχες αναφορές, όχι με τη συγκεκριμένη. Και καλό είναι να του στείλουμε και στην Επιτροπή Γεωργίας να το κοιτάξουν για αυτό το θέμα. Προς το παρόν μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνείτε? Ωραία. Καλώς, ευχαριστώ. Ξέρετε ότι είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής, μάλλον της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Και είμαι λίγο απρόθυμη να ακολουθήσω αυτό που λέτε. Αργότερα να το κάνουμε. deep into this. Να ασχοληθεί η Άγκρη αυτή τη στιγμή και κανένα άλλο. Ε, yes, we will send it up. Μάλιστα. Θα τα διαβεβάσουμε αρμοδίως και ε, στο τοπικό κτηνιατρίο ε, που είναι ε, παράρτημα του Υπουργείου Γεωργίας. Τι λέτε κύριε Κέλλη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμα αυτά που λέτε και πολύ πρακτικά και με μεγάλη κατανόηση. Σημείωσα και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν, έχουν περιορισμούς. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι όμως. Τι επιστολές θα στείλουμε στο Υπουργείο Γεωργίας στην Ιρλανδία και να τους ζητήσουμε να δείξουν κάποια ευελιξία και αν μπορούν να δώσουν τα λεφτά που χρωστάνε στον άνθρωπο. Και αν το αρνηθούν, τότε να το παραπέψουμε στην Επιτροπή Γεωργίας εδώ στο Κοινοβούλιο ή στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και τα δύο ταυτόχρονα θα γίνουν, λέει η Πρόεδρος. Ε, είναι ε, πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θα πρέπει να το κοιτάξει η Επιτροπή Γεωργίας, ό,τι και να απαντήσουν οι Ιρλανδικές Αρχές ενδεχομένως να υπάρχουν δεκάδες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι υπόψη αυτό της Επιτροπής Γεωργίας και να ασχοληθεί, να επιληφθεί. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή και ασφαλή στην Ιρλανδία και προσπαθήστε λίγο να περάσετε καλά και στις Βρυξέλλες πριν φύγετε. Now, let's move to the next. Προχωρούμε. Επόμενο θέμα, υπαρθμόν 22 ένα φορά 298 και 370. Παρευρίσκεται ο αναφερόμενος είναι ο κύριος Γιάννος Μέρη. Πού είστε? Α, εσείς είστε. Γεια σας. Ε, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή και σας δίνω το λόγο για πέντε λεπτά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα που ήρθα να σας παρουσιάσω σήμερα το βλέπουμε στον τύπο εδώ και χρόνια. Εγώ ζω στη Σλοβακία ο Ούγγρας και έχω ζήσει αυτοπροσώπως το ίδιο φαινόμενο. Πηγαίνω στον Νότιο Τυρόλο για να επισκεφθώ φίλους και σοκολάτες και μπισκότα που έχω αγοράσει στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, τα έχω πάρει μαζί μου. Και κάποια στιγμή ε, ένας φίλος μου έδωσε μια σοκολάτα της ίδιας μάρκας και γελάσαμε που έφερα το ίδιο προϊόν εγώ από την ε, Κεντρική Ευρώπη. Και δοκιμάζοντας λοιπόν τα δύο αυτά προϊόντα αντιλαμβανόμαστε ότι υπό την ίδια μάρκα το ίδιο μπισκότο έχει άλλη γεύση. Τελείως διαφορετική. Με άλλα λόγια, το μπισκότο που αγόρασα εγώ στη Σλοβακία δεν είχε ιδιαίτερη γεύση. Και όταν γύρισα σπίτι, συζήτησα με τους φίλους μου και αυτοί μου είπαν ότι και οι ίδιοι έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Ε, μετά λοιπόν από κάποια ενθάρρυνση έγραψα αυτή την αναφορά για να πιστήσω την προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Ε, ήταν η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μαθαίνει για τέτοιου είδους προβλήματα. Καλό είναι που ο Πρωθυπουργή και ο Πρόεδρος της Κομισιόν ε, ασχολούνται τώρα με αυτό το πρόβλημα. Είναι σημαντικό πιστεύω να εφαρμόζουμε τη συμμόρφωση με τους κανόνες. Ε, αναφέρθηκε ότι δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο η ποιότητα των τροφίμων. Έχουμε διαφορετική ποιότητα ε, καλλιντικών, κοσμημάτων, ε, απορριπαντικών, ε, διαφόρων ε, ειδών καθημερινής χρήσης. Απαράδεκτο. Τι συζητάμε εδώ. Λέμε ουσιαστικά ότι μια πολυεθνική εταιρεία διαθέτει το ίδιο προϊόν σε δύο αγορές διαφορετικές κρατών μελών και το προϊόν έχει άλλη ποιότητα, αποτελείται από διαφορετικά υλικά ε, σε κάθε χώρα, σε, σε, μία από τις δύο χώρες. Ε, αυτό γίνεται με πρόθεση από τον πραγωγό. Είναι μία απόφαση ε, πολιτικής παραγωγής και ας το πούμε και καθαρά. Πρόκειται για ε, επιχειρήσεις μεγάλες που σημειώνουν τεράστια κέρδη και λαμβάνουν σκεμμένα τέτοιου είδους αποφάσεις ώστε να παραπλανούν τους ε, κατοίκους ε, κρατών μελών που ε, έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα παράγοντας προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας τους εξαπατούν λοιπόν οι πολυεθνικές αυτές ενώ δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουν ορισμένους πολίτες ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας είτε είναι Ούγγροι είτε Σλοβάκοι είτε οτιδήποτε άλλο από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από το 2004. Το πρόβλημα ε, έχει ως εξή το θέμα ότι το γεγονό ότι η Επιτροπή σας ασχολείται με αυτό το θέμα ε, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει ένα εκατομμύριο ευρώ για να διερευνήσει το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ποιος θα υποπτεύσει τις σχετικές δαπάνες, ποιες θα είναι οι διαδικασίες, ποιος θα εξετάσει την όλη διαδικασία και θα την ελέγξει. Τι σας ζητάω λοιπόν, να αφήσετε την αναφορά αυτή ανοιχτή, να συνεχίσετε την παρακολούθηση των εξελίξεων και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε κάποια αποτελέσματα μαζί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω για αυτό το πρόβλημα το οποίο πλήττει εμάς, Ούγγρους, Σλοβάκους, και ουσιαστικά όλα τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 ή αργότερα. Καλή σας ημέρα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο ε, στον τομέα της εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα αυτό και για το γεγονός ότι προσωπικά ε, πραγματικά ταξιδέψατε και αναλάβετε το κόστος του ταξιδιού μέχρι τις Βρυξέλλες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα ήθελα τώρα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή γεγονός. Μέχρι 9 Ιανουαρίου τρέχοντος, ή μάλλον φέτος στις 9 Ιανουαρίου, ο Βούλγαρος διαμεσολαβητής, η κυρία Μανόλοβα μάλιστα, ε, ε υπέβαλε μια αντίστοιχη αναφορά, οπότε επειδή έχουμε τρεις αναφορές σχετικές με το θέμα, είναι παραδεκτές. Βλέπετε λοιπόν πως οι Ευρωπαίοι πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη προς τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς και θέλουμε και εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή την εμπιστοσύνη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μαρή Πολ Μπενασί. Ευχαριστώ. Uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ και για την αναφορά και για την προσωπική εμπειρία που καταθέσατε εδώ και για τα όσα παρουσιάσατε στην Επιτροπή Αναφορών. Ξέρετε και εσείς πως στην ε, ομιλία για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρσι το Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε πως δεν μπορούμε να δεχόμαστε σε κάποια τμήματα της Ευρώπης τα τρόφιμα να είναι χειρότερης ποιότητας από ό,τι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη παρόλο που οι συσκευασίε και οι, τα εμπορικά σήματα είναι τα ίδια. Λοιπόν είναι ξεκάθαρο πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πολύ σοβαρά το θέμα αυτό υπόψη και αποφάσισε να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης. Να σας πω πως το Σεπτέμβριο το σχέδιο δράσης δημοσιοποιήθηκε. Έχουμε τώρα ξεκινήσει γιατί υπάρχουν αυτά τα θέματα των προϊόντων ε, διτής ποιότητας, είναι γνωστά στην Κομισιόν εδώ και χρόνια και η δημόσια συζήτηση πέρσι το Μάρτιο έδειξε πόσο επίκαιρα είναι. Εν πάση περιπτώσει έχει πάρει η σάρκα και ο το σχέδιο δράσης και να σας πω πως καταρχήν είναι η Επίτροπος Γιούροβα υπεύθυνη για το θέμα, όπως επίσης και η Επίτροπος Μπιονκόφσκα και συζητούν με τον κλάδο των τροφίμων για το κατά πόσο υπάρχουν τέτοιου είδους πολιτικές διαφοροποιήσεις. Ζήτησαν από τον κλάδο μεγαλύτερη διαφάνεια όταν υπάρχει αυτή η πολιτική και να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με απαραίτητες προσαρμογές σε τοπικές συνθήκες, για παράδειγμα, ε, εθνικές ε, προτιμήσεις ε, και ίσως και στο λόγο της τιμής στις οποίες διατίθεται το προϊόν. Θα πρέπει οι καταναλωτές να μπορούν να κατανοήσουν αυτές τις διαφοροποιήσεις ο, ακόμα και αν αυτές τεκμηριώνονται, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση παραπλάνησης και να μην νομίζουν ότι αυτό το οποίο επιλέγουν είναι το ίδιο από χώρα σε χώρα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο δεύτερο γύρο δράσης αποφάσισε να εκδώσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές αρχές, για το πώς θα εφαρμόζουν την νομοθεσία για τα ευρωπαϊκά τρόφιμα και την προστασία του ευρωπαίου καταναλωτή και πώς θα πρέπει να αξιολογούν αυτές τις υποθέσεις κατά περίπτωση έτσι ώστε να βλέπουν ότι η πληροφορία που προσφέρεται στον καταναλωτή είναι επαρκής. Επίσης στηρίζουμε μία μεγάλη γκάμα προσπαθειών που γίνεται για ε, δοκιμή προϊόντων. Προσπαθούμε να έχουμε ε, για τη δειγματοληψία μια κοινή μεθοδολογία ένα εκατομμύριο ευρώ ε, και έχει πάει στο ε, κοινό ερευνητικό κέντρο για να διαπιστευτεί μια μεθοδολογία ε, πάντα σε συνεργασία με τον κλάδο, τους ενός καταναλωτών, τους ενδιαφερόμενους και τα εθνικά εργαστήρια. Και περιμένουμε την πρώτη μεθοδολογία να την έχουμε διαθέσιμη τον Απρίλιο και μετά θα γίνουν ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους εργαστηριακά έτσι ώστε να ε, καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα. Επίσης υπάρχουν χρήματα τα οποία έχουν ε, αποδοθεί σε ένα πειραματικό σχέδιο και κονδύλια τα οποία έχει ως σκοπό να χρησιμοποιήσει για συγχρηματοδότηση, για επιπλέον ε, δειγματοληψίες που θα γίνουν από τα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε λοιπόν πως με τον τρόπο αυτό έχουμε ένα σχέδιο δράσης το οποίο είναι πολύ γεμάτο και πως μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, πιο αντικειμενικές πληροφορίες για το εύρος του προβλήματος στον χώρο των τροφίμων και αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα γιατί βέβαια εξετάζουμε και τη δυνατότητα να το διευρύνουμε και σε άλλα προϊόντα ενδεχομένως του χρόνου. Το βασικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε το θέμα και το επόμενο βήμα είναι τα αποτελέσματα των όσων έχουμε βάλει στα σκαριά και να εξασφαλίσουμε βεβαίως πως αυτή η έλεγχη ε, και τα αποτελέσματά τους θα είναι διαθέσιμα όσο το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος από τους ευρωβουλευτές θέλει τον ε, λόγο. κύριος Γιά, ευχαριστώ πολύ τον αναφερόμενο γιατί το πρόβλημα δεν είναι νέο. Και εμείς οι βουλευτές το έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους βουλευτές από τις χώρες αυτές. Και πέρυσι αντέδρασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο έτσι κάπως ε, ελαφρύ. Είπε ότι καλά δεν βλάπτει την υγεία, είναι υγιεινά τα προϊόντα και είναι και θέμα γούστου και, και μετά άμα διαβάσεις ε, στα μικρά γράμματα, στα ψηλά γράμματα βρίσκεις και πληροφορίες αν έχεις χρόνο να το κάνεις. Αυτό είναι και η δικαιολογία για νεκά της βιομηχανίας που λέει μα τι θέλετε ε, ε, αυτό είναι θέμα συνταγής. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μείγμα θέλουμε εφόσον δεν βλάπτει τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν και τοπικές ιδιαιτερότητες, υπάρχουν κάποια μέρη που θέλουν πιο γλυκά τα μπισκότα, ξέρω εγώ, από ότι κάποια άλλη. Αυτά είναι νοησίες. βλακίες για να μην πω τίποτα χειρότερο. Γιατί εγώ όταν αγοράζω ως καταναλωτής ε, μία συγκεκριμένη μάρκα ένα εμπορικό σήμα, είτε είναι καφές, είτε είναι αναψυκτικό κόλλα, ξέρω εγώ, ε, θεωρώ ότι έχει παντού την ίδια ποιότητα. Όταν αγοράζω κοκακόλα είναι κοκακόλα. Και όταν αγοράζω κάποια περιφερειακή κάτι κόλλα, ξέρω ότι είναι άλλο πράγμα. Πολλές φορές αυτό ονομάζεται αυθαλμαπάτη, αυταπάτη, δεν ξέρω τι. Ε, αλλά δεν είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Και αν θέλετε, υπάρχουν και πιο ε, επιθετικές, ε, ξέρω πολιτικές και όταν το θέλουν υπάρχει και κοκακόλα με περισσότερη ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, δηλαδή αλλάζουν τη συνταγή και το προβάλλουν και το διαφημίζουν. Αυτό για μένα είναι εξαπάτηση του καταναλωτή και παραπλάνης. Καλό που το σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να αλλάξουν τακτική και μυαλά οι εταιρείε να έχουν τα ίδια πρότυπα ε, και τις προδιαγραφές παντού. Και όταν η σοκολάτα με φουντούκι έχει πιο πολύ φουντούκι στη Βόρεια Ευρώπη από ό,τι στη Νότια, να το γράφει επάνω. Αλλά όταν έχει μια συγκεκριμένη μάρκα, μια συγκεκριμένη γεύση, θα πρέπει να είναι παντού οι ίδιε οι προδιαγραφέ. Ευχαριστώ πολύ για την αναφορά αυτή, τον ενδιαφερόμενο και χαίρομαι που το είπε και η Κομισιόν και ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή, Ε, με εξέπληξε εμένα ευχάριστα, γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ήξη αφήξη στις απαντήσεις της. Και μόνο το γεγονός ότι άνοιξε συζήτηση μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουμε και μυαλά. Γιατί δεν υπάρχει λόγος. Η ίδια μάρκα σοκολάτα θα πρέπει να έχει την ίδια γεύση στην Ευρώπη. Εκτός αν γράφω επάνω ότι κοιτάξτε, εδώ έχω κοκακόλα με μηδέν ζάχαρη ή με περισσότερη ή με δεν ξέρω τι ζάχαρη. Αλλά ο καταναλωτής περιμένει από ε, μια μάρκα να έχει την ίδια γεύση στο προϊόν παντού. Καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και επιλαμβάνει το, θέμα του. Ευχαριστώ. Κύριε Τζίλ. Yes, Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι καινούριο αυτό. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε την σοκολάτα Cadbury's που είναι αρκετά ωραία. Δεν είμαι σίγουρος αν οι Γερμανοί τη θεωρούν σοκολάτα βέβαια, αλλά εμείς ναι. Και όταν πήγα στην Αμερική έφαγα Cadbury's και ήταν απέσια. Αλλά η ο αμερικανικός ουρανίσκος ε, τη βρίσκει μια χαρά. Είμαστε μια ήπειρος 500 εκατομμυρίων ανθρώπων με διαφορετικό τρόπο, έχουμε μεγαλώσει ο καθένα, έχουμε μάθει άλλα πράγματα, έχουμε συνηθίσει άλλα πράγματα. Πράγματα που εγώ μπορεί να θεωρώ πολύ γλυκά, άλλοι μπορεί να τα θεωρούν εντάξει. Ε, είναι θέμα ορανίσκου. Και το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι θέλουμε πλήρη εναρμόνιση, πλήρη ομογενοποίηση. Θέλουμε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ακριβώς τα ίδια προϊόντα, όπου εδώ θα νομοθετείτε τελικά και θα λέτε όταν υπάρχει μία μάρκα, τελεία και παύλα πρέπει να είναι ίδια ακριβώς σε όλη την Ευρώπη. Αλλά έτσι όμως καταστρέφεται την ελευθερία αγορά η οποία λέει ότι αν δεν σ' αρέσουν αυτά τα μπισκότα ε, σου φαίνεται ότι δεν έχουν γεύση, σταματά να τα αγοράζει. Και όταν πάβουν να τα αγοράζουν όλοι, σταματά να τα παράγει. Ή μπορεί κανεί να ζητήσει από μια εταιρεία να αλλάξει τα συστατικά. Αυτό έχει γίνει στην Βρετανία. Όταν αγόρασε, εξαγόρασε την Cadbury μια Αμερικανική εταιρεία, μετέφερε την παραγωγή ενό προϊόντο στην Πολωνία και άλλαξε η γεύση του. Οι Βρετανοί βρήκαν ότι δεν ήταν πολύ ωραία, σταμάτησαν να την αγοράζουν και χρειάστηκε να αλλάξουν και να πάνε σε άλλα συστατικά. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά, για μένα προσωπικά το ερώτημα είναι το εξή. Τι κάνουμε, αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη τη ελεύθερη αγορά, εναρμονίζουμε ολόκληρη την Ευρώπη, την κάνουμε ένα ομοιογενέ πράγμα. Δεν πιστεύω ότι θα λειτουργήσει γιατί είμαστε διαφορετικοί. Η σοκολάτα που αρέσει σε εσά είναι πιθανότατα διαφορετική από αυτή που αρέσει σε μένα. Με όλο το σεβασμό Υπάρχουν και καλύτερες χώρες όσον αφορά τη σοκολάτα, ε. Αυτό ακριβώς λέγω, ε, λέει ο κ. Τζίλς. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ που το λέτε στην ε, Βρετανία. Μας αρέσει η καντιούρη σε εσά. Ε, μπορεί να μην τη λέτε καν σοκολάτα. Εγώ είμαι Σουηδέζα και ξέρετε και η Σουηδική σοκολάτα δεν είναι και τόσο φοβερή. Δεν είναι το θέμα γαλλική ή βελγική, αλλά στους Σουηδούς αρέσει, την τρώνε. Α, καταλαβαίνω τι λέτε, λέει η Πρόεδρος, αλλά μπορώ να σας πω ότι και οι επιχειρήσεις μπορούν νόμιμα να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους για να τα προσαρμόσουν καλύτερα σε μια τοπική, ε, στα τοπικά γούστα ή στις τοπικές συνθήκες, αλλά πρέπει να το εξηγούν όμως στη συσκευασία. Και η ποιότητα πρέπει να είναι ίδια. Δεν μπορούν να βγάζουν τα καλά συστατικά και να βάζουν κα, κα, φθηνότερα συστατικά μέσα. Όταν σε μια χώρα όπως τη Βρετανία προτιμά κανείς μια σοκολάτα πιο, με πιο μαλακή γεύση, με πιο γλυκιά γεύση, ε, θα πούνε ωραία παίρνουμε μια γαλλική μάρκα υψηλής ποιότητας ε, αλλά εξηγούμε ότι την έχουμε προσαρμόσει στις απαιτήσει ε, των Βρετανών. Αυτό είναι θεμητό. Σύμφωνα με την νομοθεσία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να υποβαθμίζει την ποιότητα. Δεν είναι διαπραγματεύσιμη η ποιότητα. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Τζίλους. Αυτό που λέω, δεν θέλουμε απάτη, δεν θέλουμε εξαπάτηση των καταναλωτών. Και εκεί έρχεται η επισήμανση. Πέτερ. Ήθελα μόνο ε, να δω ε, τι κάνουν οι εταιρείες. Στην πύρα, ας πούμε. Έχουμε εταιρείε που διευρύνονται, που έχουν εξαγοράσει ε, μικρές ειδοποιίες και βγάζουν 50 είδη μπύρας. Το γράφουν όμως. Ποια είναι η διαφορά. Ε, υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες γεύσης για το ζήθο, αλλά το λένε. Ε, δεν έχουν σκεφτεί ποτέ να κάνουν μια ενιαία μπύρα για όλη την Ευρώπη με διαφορετικές συνταγές κάθε φορά. Λοιπόν, όταν έχει μια μάρκα, θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η ίδια ποιότητα. Και αν υπάρχουν τοπικέ ιδιαιτερότητε που υπάρχουν, γιατί ισχύει αυτό στη ζωή, θα πρέπει να έχω ε, ε, μια επιθετική διαφάνεια, δηλαδή να το προβάλλω. Αυτό ε, δεν θα πρέπει να τρέχω στο ίντερνετ να το βρω, να δω τι σιρόπι έχει μελάσα ή ζάχαρη, να το γράφει πάνω το προϊόν. Ακριβώς την πείρα είναι το αντιπαράδειγμα. Δεν θα τολμούσε ποτέ κανείς να φτιάξει μια ενιαία συνταγή μπύρας για όλη την Ευρώπη και με το ίδιο όνομα. Πώς να το πω δηλαδή. Καμιά φορά επαναπαύονται και οι εταιρείε ε, αξιοποιούν, εκμεταλλεύονται τη φύρμα, το όνομά του στο εμπορικό σήμα χωρίς διαφάνεια. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, να το λένε αυτό, να το δηλώνουν. Πρέπει να σας πω ότι το συζήτησα και με τις εταιρείε. που και αυτοί έτσι με υπεκφυγές απάντησαν, δεν μπήκαν ποτέ με ειλικρίνεια στη συζήτηση και παρακαλώ να το λέει κάπου, ξέρω εγώ, Coca-Cola made in Hungary ή made in Norway, να μην λέμε ότι είναι η ίδια Coca-Cola παντού. Γιατί αν δεν υπάρχει με διαφάνεια σήμανση γεννάται υποψία, υποψία ότι είναι ίσονος ε, ποιότητας, χαμηλότερης και μεγαλύτερα τα κέρδη. Ενώ στην πύρα βγαίνουν και το λένε. Γιατί δεν το κάνουν όπως στην πύρα. Ότι ορίστε ποια η συνταγή επάνω Στη Τσεχία ούτε ξέρω πόσα είδη μπύρας υπάρχουν. Δηλαδή ήδη από το όνομα καταλαβαίνεις ποια είναι η συνταγή. Στην Coca-Cola γίνεται το αντίθετο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση φαντάζομαι, αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηκώνει το δάχτυλο και λέει «Παιδιά, για ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε τι κάνετε εδώ πέρα». Ωραία. Να παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα, παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Ευχαριστώ. Κύριος Τσάκη. Ε, όσον αφορά τη θέση του Πέτερ Γιάρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε σαφέστατα ότι αυτό είναι πρόβλημα πράγματι και ότι απαιτείται δράση. Αγαπητοί συνάδελφε, μία πρόταση. Χρειαζόμαστε σαφεί κανόνε στο παιχνίδι αυτό. Δίκαια πράγματα. Καλό θα είναι λοιπόν να την κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά, να συνεχίσουμε το διάλογό μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε τι θα γίνει. Χρειαζόμαστε μια σαφή δίκαιη κατάσταση. Ε, Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μέρη, θέλετε να ξαναπάρτε το λόγο, να απαντήσετε στο όσο ακούσαμε. Ναι. Ευχαριστώ. Στα αγγλικά θα μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να λησμονούμε και να συγχαίουμε. Εγώ δεν μιλάω για εμπορικά σήματα, μάρκες. Αλλά, ούτε να αναφέρω μάρκα, αλλά όταν αγοράζω μια σοκολάτα κάπου στην Ευρώπη που έχει ένα συγκεκριμένο εμπορικό σήμα, μια μάρκα, θα πρέπει παντού αυτή να έχει την ίδια σύνθεση. Εμείς δεν θέλουμε αρμονισμένα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη, αλλά όταν έχει μια συγκεκριμένη μάρκα που πουλάει κάτι γνωστό και όλοι γνωρίζουν ε, ότι παντού ε, κυκλοφορεί το ίδιο προϊόν, και έχει την ίδια γεύση, αυτό αναζητούμε. Οι περισσότεροι από εμά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον στην Ανατολική Ευρώπη, μάθαμε τα προϊόντα αυτά από ταξίδια στη Δυτική Ευρώπη ε, μετά τη μεταπολίτευση και γινώντας ε, στα σπίτια μας ξαφνικά άρχισαν να πουλάνε ίδιες μάρκες τα προϊόντα τους στην Ουγγαρία ας πούμε και δεν ήταν ίδια γεύση. Αυτό θέλω να πω, να το προσέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ και να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μας. Και δεν θα πρέπει να μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ζούμε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το αντίθετο, χάρη στην Ευρώπη, λέει η Πρόεδρος, μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα διατηρηθεί η ποιότητα. Ωραία. Νομίζω αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα, να αφήσουμε ανοιχτή φυσικά την αναφορά και να περιμένουμε το κοινό ερευνητικό κέντρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βγάλει μια κοινή μέθοδο. Πότε είπατε τον Απρίλιο, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της Άνοιξης φέτος και μετά να έχουμε τα στοιχεία και τις ακράδαντες αποδείξεις που χρειαζόμαστε ε, μετά από τα όσα ανέφερε ε, ο αναφερόμενο μας. Καλό θα ήταν, κύριος Μέρη, να στείλουμε και στις ε, σλοβακικές αρχές και στις ουγγρικές την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία τους ε, μια επιστολή να πούμε πώς ανησυχούν οι πολίτες και πώς θέλουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές. Αυτές οι δύο αναφορές θα πρέπει να παραμείνουν ενωμένες. Υπάρχει και μια τρίτη που επίκειται, γιατί μου κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες τον Ιανουάριο. Λοιπόν, παράλληλα να τα εξτάσουμε αυτά τα θέματα και να προσπαθήσουμε να τους επιφυλάξουμε την ίδια μεταχείριση. Συμφωνείτε? Ωραία. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε. Χαιρετισμό στη Σλοβακία όταν γυρίσετε. Προς το παρόν φάτε και καμιά βελγική σοκολάτα πριν φύγετε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο σημείο, που είναι η αναφορά υπαριθμό 15 για την εναρμόνιση των παραμέτρων ασφάλισης για την αποζημίωση ζημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το σημείο 23 της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την αναφέρουσα, που είναι η κυρία Μογνώτσα, που προσωπεί τον αναφέροντα και σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά. Αγαπητοί κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί όσοι είστε εδώ. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κωνσταντζά Σκεράσα Μουνιώτσα και είμαι η αδερφή της Ελίζας, μια 25χρονη ε, φοιτήτρια που έχασε τη ζωή της στη Βαρκελόνη όπου είχε πάει για ένα Εράσμους ένα ταξίδι που είχε οργανωθεί από την Ισπανική Οργάνωση Εράσμους Student Network στις 20 Μαρτίου του 2016 πριν δύο χρόνια έχασαν ε, τη ζωή τους 13 ε, φοιτήτριε, 6 7 Ιταλίδες και 6 από διάφορες υπηκότητες. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το δυστυχές συμβάν όπου έχασαν τη ζωή τους 13 ε, νεαρές ε, κοπέλες πολίτες της Ευρώπης που συμμετείχαν στο Εράσμο στο οποίο συμμετέχουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες νέοι φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Ήθελα να προσθέσω ενημερωτικά ότι ακόμα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το δράμα. Μετά από δύο χρόνια δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες της Ισπανίας και δεν έχουν ε, βρεθεί ε, ενοχή ούτε υπεύθυνοι. Οι Ισπανοί δικαστέ έχουν αρχιθετεί στην υπόθεση θεωρώντα ότι δεν υπάρχει υπεύθυνο παρότι ήταν σαφή η ευθύνη του οδηγού. Δύο χρόνια μετά από το τραγικό συμβάν και τι προσφυγέ των οικογενειών δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη ακόμα. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω εξ ονόματο τη Διεθνού Ένωση Γονεί τη Γενιά του Εράσμου, ενωμένοι ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό που συστήθηκε από γονεί ε, ε, κοριτσιών στην Καταλωνία με την αναφορά 0015-2017 για την εναρμόνιση των παραμέτρων ασφάλισης για την αποζημίωση ζημιών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσιάστηκε από τον κύριο Σιμών Βεράλτη. Θα ήθελα να ε, επιστήσω την προσοχή σας στην διαφοροποίηση και στα κενά και στις διαφορές που υπάρχουν από τις διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Έχουμε τον κανονισμό Ρώμα 2 και την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C550 του 2015. Δεν θα τις αναλύσω εδώ, αλλά θέλω να σας αναφέρω τι συνέβη σε εμά. Δεδομένη τη σημερινή ευρωπαϊκή νομοθεσία και βάσει των όσων προβλέπονται από την απόφαση C350 του 2015, Καταλήγουμε στο ε, παράλογο συμπέρασμα ότι οι συγγενείς ε, των ε, κοριτσιών από την Ιταλία που έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία μπορούσαν να αποζημιωθούν βάσει των ισπανικών κανόνων τρεις ή τέσσερις φορές λιγότερο από αυτό που θα δικαιούνταν στην Ιταλία, αν είχε συμβεί το ατύχημα στην Ιταλία. Αντιστρόφως, εάν οι Ισπανίδες κοπέλες είχαν ένα τέτοιο ατύχημα στην Ιταλία, οι οικογένειές τους θα είχαν αποζημιωθεί τριπλάσια, τετραπλάσια από ότι θα, αυτό που θα συνέβαινε στη χώρα τους. Επιπλέον, ε, σε χώρες ε, ευρωπαϊκές όπως η Ισπανία, αντίθετα την Ιταλία, τα νομικά έξοδα τα καταβάλουν ε, οι ενάγοντες. Αν, ανεξάρτητα από την απόφαση. Είναι σαφές λοιπόν ότι είναι άδικο το σημερινό σύστημα Συνεπώς σας ρωτώ, η ζωή ενός Ευρωπαίου πολίτη δεν πρέπει να έχει την ίδια αξία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτή την αρχή θα έπρεπε να αγωνίζεται η Ευρώπη, να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει μια εναρμόνιση των ασφαλίσεων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τουλάχιστον οι συγγενείς των θυμάτων ατυχημάτων στο εξωτερικό να αποζημιώνονται βάσει των κανόνων των χωρών όπου ζούσαν ε, το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής τους στα θύματα. Αυτό προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών που κάθε χρόνο ε, ε, περνούν τα σύνορα των κρατών μελών για εργασία, σπουδές ή διακοπές. Φυσικά ε, κανένα ναι, υλικό μέσο δεν θα μας ε, επιστρέψει τα κορίτσια μας αυτά, αλλά επειδή μιλάμε εδώ για τη γενιά Εράσμους, θεωρούμε ότι πρέπει να φροντίσουμε να μην ξαναγίνουν παρόμοια συμβάντα, ώστε οι νέοι Ευρωπαίοι που θέλουν να ακολουθήσουν τα χνάρια της αδερφής μου της Ελίζα και άλλων ε, νεαρών κοριτσιών από όλες τις χώρες, να ε, απολάβουν καλύτερων εγγύσεων ε, καθημερινά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Καλύτερη ασφάλεια ταξιδιών και ε, μέσων συγκοινωνιών, καλύτερες οδικές υποδομές, πιο σαφή κανόνες ασφάλισης και αποζημίωσης. Ήθελα να υπενθυμίσω το κοινοβουλευτικό ερώτημα που πρόθεσαν η κυρία Σιλβία Κώστα και ο Μίχαλ Κράμερ σε σχέση με τα κριτήρια ε, προστασίας των φοιτητών Εράσμους. Το πρόγραμμα Εράσμους ε, θέλει να δημιουργήσει τους νέους Ευρωπαίους πολίτες. Έτσι λοιπόν μας φαίνεται αδιανόητο ότι σήμερα νέοι μπορεί να ε, μην έχουν μια υποχρεωτική ασφάλιση και αποζημίωση σε περίπτωση ατυχημάτων. Και σε τέτοια δραματικά ατυχήματα όπως αυτά που έβληξαν τις δικές μας ε, κοπαέλες και τους άλλους φοιτητές δεν αποζημιώνονται δίκαια. Πρέπει λοιπόν πέραν από τους κανόνες αποζημίωσης το πρόγραμμα Εράσμους να προβλέπει την υποχρέωση να καλύπτονται από επαρκή ασφαλιστικά συμβόλαια οι φοιτητές όχι μόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα πανεπιστήμια αλλά και σε όλη του τη διαμονή σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι νομοθεσίες, οι πληροφορίες που δίδονται στους νέους φοιτητέ ε, δεν είναι σαφείς. Επίσης, ε, ασαφείς είναι και οι ευθύνες των πανεπιστημίων, τα οποία υποδέχονται τους φοιτητέ και των ενώσεων που συνδέονται με αυτά τα πανεπιστήμια και τα οποία οργανώνουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Ένα πρώτο βήμα ρεαλιστικό θα ήταν η διασφάλιση ίσων προτύπων στα ασφαλιστικά συμβόλαια που ε, διαθέτουν τα διάφορα πανεπιστήμια στο πλαίσιο των προγραμμάτων Εράσμους. Επίσης πρέπει να εμβαθύνουμε τη λειτουργία εντός του προγράμματος Εράσμους μη κερδοσκόπων οργανισμών που λαμβάνουν ενωσιακά κονδύλια όπως η ECN να γίνουν έλεγχοι όσον αφορά τη χρήση των κονδυλίων που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το πόσο χρησιμοποιούνται σωστά. Κάποιες τέτοιες ενώσεις συχνά λειτουργούν ως πρακτορία ταξιδίων χωρίς να έχουν τις ικανότητες ε, και χωρίς να προσφέρουν την ασφάλεια που απαιτείται, ούτε τις εγγύησεις. Ε, στην περίπτωση των δικών μας κοριτσιών, σε αυτό το τραϊκό ε, ταξίδι που οργανώθηκε από την ESN της Ισπανίας από τη Βαρκελόνη μέχρι τη Βαλένθια στο πλαίσιο ενός προγραμματός Εράσμους. Ο ίδιος ο οργανισμός, ο ESN, ε, αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για το συμβάν και η διεθνής ESN των Βρυξελών ε, λέει ότι ευθύνονται οι τοπικές αρχές, οι τοπικές ενώσεις. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Είμαι βέβαιη ότι στο μέλλον θα υιοθετήσετε όλα τα νομοθετικά μέτρα και τεχνικά και διοικητικά μέτρα τα οποία απαιτούνται ώστε τα παιδιά των διαφόρων χρόνων να μπορούν να μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν να είχαν ένα κοινό σπίτι με επαρκείς παρόμοιες εγγύσεις για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για το θάρρος σας να ταξιδέψετε εδώ για να έρθετε να μας διαφωτίσετε για το θέματα αυτά. Επιτρέψτε μου επίσης εκ μέρους της ε, Κομισιόν να σας εκφράσω τα βαθιά μας ελληπιτήρια για την απώλεια της αδερφής σας. Ήταν πραγματικά πολύ θαραλέο από πλευρά σας να έρθετε εδώ και να μοιραστείτε μαζί την ε, ιστορία σας. Θα καλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο στα πλαίσια των όσων μόλις ακούστηκαν. Έχω εδώ ε, τον κύριο Λύση Καλησπέρα σας. Λυπάμαι πάρα πολύ που άκουσα αυτή την τόσο συγκινητική ιστορία και είμαι στην πολύ δύσκολη θέση που θα κληθώ να εξηγήσω το ποια είναι η νομοθετική θέση και ως εισαγωγή να σας πω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την οδηγία για τις ασφαλίσεις, το τι γίνεται, το τι δεν γίνεται και θα προσπαθήσω ε, να δω όλες τις ε, πλευρές να σας πω πως η οδηγία αυτή έχουμε το σύστημα της πράσινης κάρτας που είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό ασφάλισης και που επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να ταξιδεύουν διασυνοριακά χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν ε, ασφάλιση αλλοδαπής. Αυτό το σύστημα με την πράσινη κάρτα δίνει τη δυνατότητα σε περίπτωση ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα σε άλλο κράτος μέλος ε, με ε, αλλοδαπούς οδηγούς να πληρώνει κάποιες αποζημιώσεις. Τώρα έχουμε αναβαθμίσει το σύστημα αυτό και πρέπει να σας πω πως προσφέρει για παράδειγμα ελάχιστα επίπεδα κάλυψης Και θα πρέπει αυτά τα ασφαλιστήρια να καλύπτουν για παράδειγμα και τις ε, ζημίες, τις και την ε, ε, σωματική βλάβη. Αυτό δεν σημαίνει συμβαίνει με την ε, πράσινη κάρτα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε τι γίνεται με την κάλυψη των πεζών και των ποδηλατών. Αλλά πρέπει να σας πω με τις αποζημιώσεις δεν είμαστε απολύτως σίγουροι τι συμβαίνει γιατί είναι κάτι διαφορετικό και για να κλείσω την περιγραφή της οδηγίας έχουμε για τα θύματα επισκέπτες που νομίζω είναι η περίπτωση που συζητάμε Δεν ξέρω αν ήσασταν παλαιότερα, ήταν παλαιότερα το θύμα και κάτοικο στην Ισπανία, αλλά στην περίπτωση αυτή γίνεται η, δυνατή η αίτηση αποζημίωσης για όλους όσους έχουν υποστεί βλάβη. Τώρα, για την αποζημίωση την ίδια, για την αποζημίωση, λοιπόν, για τα θύματα επισκέπτες, στη μελέτη που ζητήσαμε, ε, εντοπίσαμε πως υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε επίπεδο αποζημίωσης Και να σας πω πως τα διαφορετικά κράτη-μέλη ήταν διαφορετικά για επίπεδα αποζημιώσεις. Γιατί, για παράδειγμα, είναι διαφορετικό το επίπεδο ιατρικών δαπανών. Άλλο αν έχει τραυματιστεί, ε, άλλο αν ε, το αστικό δίκαιο σε καλύπτει ε, και, για παράδειγμα, σε κάποια κράτη-μέλη δεν δίδεται καθόλου αποζημίωση για περίπτωση ψυχολογικής βλάβης. έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη σε κάθε κράτος μέλος, έχει να κάνει με την απώλεια δυνητικού εισοδήματος, οπότε η κατάσταση είναι αυτή και τα όσα κλείσανε το 2008 ήταν το εξή πως ότι το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι τόσο τεράστιο. Βεβαίως δεν μπορούμε τραγικές υποθέσεις σαν αυτή την οποία ε, περιγράφεται δεν μπορούμε να τις ε, σπρώξουμε στην άκρη, αλλά η μελέτη του 2008 δεν εντόπισε μεγάλο πρόβλημα με τέτοιου είδους υποθέσεις. Δηλαδή, μάλλον μέσω αναλογικότητας και επικουρικότητας το θέμα αυτό πρέπει να αφαιθεί στο τρέχον σύστημα. Δυστυχώς, λοιπόν, αυτά έχω να απαντήσω. Δεν σχεδιάζουμε να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο συγκεκριμένα για το θέμα αυτό και είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζω, που αντιμετωπίζω τέτοιου είδους ε, καταγγελία στα τέσσερα χρόνια που ασχολούμαι. Και δεν μπορώ εγώ βέβαια να προτείνω κάποιο τρόπο δράσης, ούτε έχω εντολή για να κάνω κάτι τέτοιο. The floor is open Λοιπόν, συνάδελφοι, ανοίγει η συζήτηση. Ο Πέτερ Λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι ότι ο Έρεσμος ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο σχέδιο, success story. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ευτυχώς θα πω εγώ. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν πάντα τραγικά ε, περιστατικά, αλλά φυσικά είναι τραγικό όταν κάποιο έχει νεκρό στην οικογένεια και μετά δεν μπορεί να βρει και το δίκιο του και να αποζημιωθεί. Αυτό επιτείνει μετά το αίσθημα ε, της ατιμορρησίας και της αδικίας. Γιατί σου λέει ε, εγώ ασφαλίζομαι ε, για πάνε ενδεχόμενο, για να μην συμβεί κάτι. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάτι για να αποτρέψει κάτι άλλο. Ή δεν το επιδιώκει, αλλά σε περίπτωση που συμβεί κάτι να υπάρχει δικαιοσύνη. Και ρωτώ τους συναδέλφους, γιατί εγώ δεν σκαμπάζω απονομικά, ε, στο Εράσμους ε, μπορούμε να προβλέψουμε καμία ασφάλεια που να ασφαλίζει ε, τους φοιτητές που ζουν στο εξωτερικό. Όταν πάω εγώ ταξίδι, το πρώτο πράγμα ε, που κοιτάω δεν είναι να αποζημιωθεί κάποιος αν στη τη ζωή μου γιατί υποθέτω θα γυρίσω υγιής. Αλλά επειδή ως πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύεις ε, και ε, είσαι σε μια άλλη χώρα και σου συμβεί κάτι, δεν μπορεί να υφίστασει αδικίες. Γιατί δεν το κάνουμε και στον έρασμο να προβλέψουμε μια ασφάλεια για τους φοιτητές ή στα άλλα προγράμματα. Να προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή ασφάλεια που να προβλέπει δίκαιη αποζημίωση και να μην κοιτάω κάθε φορά που έγινε το δυστύχημα στα σύνορα, από ποια πλευρά των σύνορων, ποιο έφταιγε. Είχε γεννηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάποιο κράτος μέλος. Αυτά όλα είναι δυσάρεστα και στενάχωρα πράγματα. Αυτό θα ρωτούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συναδέλφους. Μπορούμε στον έρασμο να βάλουμε ένα σύστημα ασφάλειας. Γιατί μπορεί να είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά είναι τραγικά και δεν θέλουμε να υπάρχουν. Ευχαριστούμε, Πέιτερ. Και τώρα στρέφομαι στη Σιλβία Κώστα, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι μια από τις πρώτες φορές που είστε εδώ στην Επιτροπή μας. Σας καλωσορίζω θερμά. Έχουμε δουλέψει μαζί πολλές φορές ε, στην Κάλτε, οπότε χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και εγώ ε, ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το τρομακτικό δυστύχημα γιατί με έχει συγκινήσει πολύ. Ευχαριστώ, θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Ήθελα να πω και εγώ ευχαριστώ στην Κωνσταντζα ε, στην Κωνσταντζα Σκαρασαμουνιώτσα για το τεράστιο θάρρος της και για την ακρίβεια και τη σαφήνεια με την οποία παρουσίασε αυτό το γεγονός. Εγώ ήθελα να πω ότι γνωρίζω την οικογένεια, τις οικογένειες πολλών από αυτά τα κορίτσια από την Ιταλία. Είχαμε και την τιμή να φυτέψουμε κάποια δέντρα στη Ρώμη σε ένα μεγάλο πάρκο με τους γονείς οι οποίοι είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, δημιούργησαν αυτή την ένωση για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο για το μέλλον, για τα άλλα παιδιά. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Θεωρώ ότι εδώ έχουμε τρία προβλήματα. Το πρώτο, και εγώ το λέω ως άνθρωπος από την Επιτροπή Πολιτισμού, είναι κάτι για το οποίο εγώ έχω ζητήσει από την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδείας να επαληθεύσει κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω όσον αφορά τις εγγυήσεις, τα ασφαλείς αυτές των παιδιών που φεύγουν σε εράσμους. Ποιο είναι το πρόβλημα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ε, στέλνονται από τα προεπιστήμια και αναφερόμενα στους κανόνες που υπάρχουν στην κάθε χώρα. Ε, οπότε η Κωνστάτσα καλυπτόταν από τους κανόνες τους Ισπανικούς. Αυτή είναι μία πτυχή. Η πράγματι αποζημίωση θα ήταν τριπλάσια αν ήταν στην Ιταλία. Οπότε όχι μόνο χάνουμε μια ζωή που δεν μπορεί να επιτρέψει η Ευρώπη, αλλά και τα χρήματα. Δεύτερον, στο κομμάτι του ασφαλιστηρίου συμβολέου λέμε, αναφέρομαστε στα πράγματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα Εράσμους, αυστηρά. Αλλά ξέρουμε ότι το πρόγραμμα Εράσμους είναι και ένα πρόγραμμα ε, ιδιότητας του πολίτη, γνωριμίας. Ε, έκανα μια εκδρομή δηλαδή για να γνωρίσουν τα κορίτσια τη χώρα μέσω του ESN που είναι μια ένωση, μια χαρά. Αξιοπροπέστατη αποτελεί κομμάτι του ευρωπαϊκού δικτύου που υποστηρίζεται και από την Κομισιόν και προσφέρει καλόπιστα σίγουρα τέτοιου είδους ε, εκδρομές, επισκέψεις, ε, πρωτοβουλίες, ε, ένα νυχτερινό ταξίδι ολονύκτιο με επιστροφή το πρωί. Εδώ το θέμα δεν ήταν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια, το λέω ειλικρινά. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει η Γενική Διευθύνση Παιδεία και Πολιτισμού να δώσει κατευθυντέ γραμμέ στα σχετικά δίκτυα που υποδέχονται φοιτητέ, ώστε να εφαρμόζουν κριτήρια τέτοια που να υποδέχονται και να προσφέρουν ευκαιρίε ε, στου φοιτητέ αυτού ε, πέραν ε, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με κάποιε εγγύησει. Το τρίτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα τη πολιτική, τη εναρμόνιση. Εγώ έχω δει τη μελέτη του 2008 αλλά το 2008 είναι ξεπερασμένο πια. Εκεί αναφερόταν ότι τέτοιου είδου καταστάσεις ε, δεν εμφανίζονται συχνά ε, τόσο κρίσιμες καταστάσεις έλλειψης εναρμόνισης των πολιτικών. Ε, πιστεύω ότι για κάποια στάνταρ θα μπορούσαμε να έχουμε όμοια, τουλάχιστον σε περιπτώσεις σοβαρές, όπου χάνεται κάποια ζωή χωρίς μεγάλε επιπτώσεις για την εσωτερική αγορά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα. Γιατί ε, ξέρετε, είναι μεγάλη η επιρροή. Έχουμε χάνονται ζωέ. Και δεύτερον, διότι πιστεύω ότι καθώς αυξάνεται η διεθνής κινητικότητα και χάρη στο Εράσμους έχουμε είναι πολλοί που επωφελούνται από την κινητικότητα και εκεί έχει μια ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να περάσει, να κάνει ένα πρώτο βήμα βάσει αυτών των νέων ώστε να καταλήξουμε να συζητάμε για εναρμόνιση των ασφαλιστηρίων συμβολέων τουλάχιστον για κάποιε ιδιαίτερε περιπτώσει, τι πιο σοβαρέ και για κάποια κοινά στάνταρ. Σε αυτό προσθέτεται ότι δυστυχώ η Ισπανία ακόμη δεν έχει συνάψει μετά από διάφορε διαδικασίε, δεν έχει καταλήξει κάποιο συμπέρασμα του ποιο είναι ο υπεύθυνο, ποιο είναι ο ένοχο. και δεν έχει δοθεί καμία ικανοποίηση στι οικογένειε αυτέ. Οι οικογένειε αυτέ ε, ε τι έχουν ορίσει κάποιε από αυτέ. Δεν έχουν τα μέσα. Είναι απαράδεκτο να υφίστανται τέτοια, ε, τέτοια μεταχείριση, άνηση. Οπότε θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να μην την κλείσουμε, να θεωρήσουμε ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη. Όχι μόνο στο πλαίσιο του Εράσμου. Εγώ έχω ζητήσει και στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων να γίνουν διευκρινήσει γι' αυτό και να αρχίσουμε να καθορίζουμε μία πρώτη αρχή ε, ασφαλιστήριο συμβολέων που να διασφαλίζουν την καλή ζωή, την καλή μεταχείριση, την επιβίωση δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση ε, παιδιών που έρχονται από όλες αυτές τις χώρες. Αυτό θα είναι απέτηση των νέων γενναίων στην Ευρώπη και εμείς θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη ενώπιον τους. Ευχαριστώ. Thank you so much. And I believe... Ευχαριστώ πολύ και πολλοί από εμά εδώ είτε ήμασταν οι ίδιοι φοιτητέ με τον Εράσμους. Εγώ πέρσι έστειλα το γιο μου στην Γαλλία, ευτυχώ έχει επιστρέψει τώρα στην ε, Σουηδία, αλλά δεν τα σκέφτεσαι τα πράγματα ότι θα σημούν στο παιδί σου όταν το στέλνει δέχεσαι ότι θα το δεχτεί ένα πολύ ε, καλό πανεπιστήμιο, αλλά δεν σου περνάει ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να συμβεί τέτοιο πράγμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να λυθούν. Ε, παράλληλα, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Εράσμο, ήταν πρωτοπόρο και θα πρέπει να βρούμε και πρωτοπόρο λύση τώρα. Ο κύριος Τζιλ, ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό. Και δυστυχώς, μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία τέτοια περίπτωση γιατί όσο προχωράει ο καιρός αυξάνονται οι πιθανότητες ε, δυστυχημάτων και θανάτων. Χρειάζεται μια λύση μακροπρόθεσμη και για τις οικογένειες θα πρέπει ε, ε, να τους βοηθήσουμε να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο να πενθήσουν και να προχωρήσουν. Ε, στην Ισπανία δεν μπορεί να δοθεί προτεραιότητα ε, στη δικαιοσύνη σε αυτό το θέμα για να μάθουν οι οικογένειες πραγματικά τι έγινε και να πάνε παρακάτω. Και κάτι άλλο. Μια οικογένεια από τη Ρουμανία, ξέρω εγώ, ε, ε, δεν είναι το ίδιο για την οικογένεια αυτή 1000 ευρώ με μια οικογένεια από τη Γαλλία ή το Βέλγιο. Έχουν διαφορετική αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Άρα εγώ θα ήθελα ε, μια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να λέει ότι ανάλογα με την καταγωγή της χώρας η μέγιστη αποζημίωση είναι τόσο. Είναι από την Ιταλία, από την Ισπανία κτλ. και να πάρουν την υψηλότερη αποζημίωση. Αυτό νομίζω είναι μια λογική λύση. Δυστυχώ η λογική δεν πριτανεύει πάντα. Κύριε Σκοτσολίνο. Ε, Φαίνεται υπερβολικό τώρα να κάνει κανεί σχόλια περί το πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να επικαιροποιήσει τη μελέτη του 2008. Είναι προφανές. Είμαστε το 2018, έχουν περάσει 10 χρόνια και στο μεταξύ. Ε, έχουμε τεράστια αύξηση των Εράσμου. Εμείς μάλιστα επιμένουμε να διευρυνθεί η συμμετοχή των νέων στο Εράσμους. Και γνωρίζουμε ότι το θέμα της κινητικότητα πλέον υπάρχει, δεν είναι ότι πάει κανεί σε ένα πανεπιστήμιο και μένει εκεί. Πολύ συχνά ε, το πανεπιστήμιο ε, χρησιμοποιείται ως πύλη για να πάει κανείς αλλού και δυστυχώς ε, είχαμε αυτά τα κορίτσια που υπέτσαν ε, αυτή την άτυχη συγκυρία. Θα πρέπει να επικαιροποιηθεί λοιπόν ε, η μελέτη του 2008. Αυτό πρέπει να απαιτήσουμε από την Κομισιόν. Και μετά θα δούμε τι λύσεις μπορούμε να βρούμε και εμείς έχουμε το καθήκον να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά έως ότου λάβουμε ουσιώδεις απαντήσεις από πλευράς κομισιών και όσον αφορά αυτή την επικαιροποίηση μου φαίνεται προφανές ότι το να έχουμε αυτή τη στιγμή ως σημείο αναφορά σε ένα κείμενο του 2008 ε, δεν έχει νόημα δεδομένης της ε, ε, τεράστιας αύξησης των φοιτητών Εράσμους και της ανεπαρκούς νομοθεσίας από αυτού του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν να σας ξαναδώσω το λόγο κυρία Σκαράσα Μουνιώτσα. Δύσκολο να το προφέρω το όνομά σας. Σας ευχαριστώ όλους. Και κατά τη δική μου απόψη η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που ε, είναι το 2008 πρέπει να επικαιροποιηθεί. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στις περιπτώσεις που Ευρωπαίοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους, αλλά και σε περιπτώσεις όπου, όπως έχει συμβεί στη δική μας περίπτωση, να υπάρχουν πολλοί φοιτητέ που να έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες. Μου φαίνεται περίεργο λοιπόν ότι είναι τόσο λίγε περιπτώσει δεδομένου ότι ταξιδεύει πολλοί κόσμο. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Εράσμο, αναφέρομαι στα ταξίδια από τη μια χώρα στην άλλη. Μου φαίνεται παράλογο να μην υπάρχουν περιπτώσει ε, με ατυχήματα. Ε, ατυχήματα σε Ευρωπαίου πολίτες που ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ λοιπόν ειλικρινά για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε σας. Λοιπόν, να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα θα ήθελα μετά από τη συζήτηση αυτή. Όπως μπορεί να θυμάστε, παρόλο που ο χρόνος περνάει γρήγορα, τον Ιούλιο του 2017 είχαμε ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ακριβώς για αυτό το θέμα. Από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραθέτω λίγο να αναλάβει να ορίσει ε, ελάχιστους κανόνες πανευρωπαϊκά έτσι ώστε να μην χάνουν τα δικαιώματά τους ε, σε αποζημίωση εκείνοι που ενέχονται σε ε, τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα σε άλλη χώρα. Βεβαίως θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να στείλουμε τη δεκμήριωση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Γιούρι ως παράδειγμα πραγματικού περιστατικού ε, που αντιστοιχεί στο ψήφισμά τους του Ιουλίου και να τους ζητήσουμε να κοιτάξουν ε, τι συνέχεια μπορεί να δοθεί στο πλαίσιο του ψηφίσματος. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε στην Επιτροπή Μεταφορών ενημερωτικά και στην Επιτροπή Πολιτισμού. Πολιτισμού βεβαίως, γιατί το Εράσμος υπάγεται εκεί. Και προσωπικά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή αναπτύσσεται το πρόγραμμα Εράσμος, όλο αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε, της ασφάλισης, παράλληλα. Αν γίνεται, δεν ξέρω. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να το ψάξει η Επιτροπή Πολιτισμού. That we also take... Όντως, και θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό που επανέλαβαν πολλοί συνάδελφοι η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ηλικίας 10 ετών. Και αν έχουν συμβεί πράγματα μέσα σε 10 χρόνια, μπορείτε να φανταστείτε πόσα θα συμβούν μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οπότε να το κοιτάξουμε αυτό σοβαρά παρακαλώ. Και με βάση κάποιες προσωπικές τραγωδίες. Ξέρουμε υπάρχει ένα σύστημα συλλογικής αποζημίωσης, συλλογικών αγωγών κτλ. Αυτό το συζητάμε, αλλά δεν είναι διασυνοριακό. Και αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Θα ήταν ε, χρήσιμο. Αυτό προτείνω για να προχωρήσουμε. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θα το διαβεβάσω αρμοδίως. Να το διαβιβάσετε παρακαλώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ξέρετε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη διοργανική συνεργασία και είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για να βρούμε μια λύση αποδεκτή. Και ενημερωμένοι στην Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν υφίστανται πλέον ή δεν είναι τύχη. Προσπαθούμε να, να γρεμίσουμε αυτά τα τύχη και να βρούμε κοινέ λύσεις. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Μια φορά και έναν καιρό ήταν το Εράσμος πρωτοπόρο πρόγραμμα. Ε, τώρα είναι μεγάλη προτεραιότητα να βρούμε μια λύση. Καλή σας τύχη και καλή μας τύχη εδώ στο Κοινοβούλιο και σε εσά που ήρθατε από τόσο μακριά από την Ιταλία να μας παρουσιάσετε την αναφορά σας. Ευχαριστώ και πάλι και να διαβιβάσετε χαιρετισμού στους φίλους και την οικογένειά σας. Now, let's move to the presentation of another study. Προχωρούμε. Παρουσίαση άλλης μελέτης με τίτλο «Αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη». Παρευρίσκεται η Μαρτίνα Wait a minute. Okay. We have the expert with us. Α, έχουμε την Άφηρα Μάσον που είναι η Διευθύντρια του Έργου και Νομική Σύμβουλος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα βασικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης που έγινε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και να σας πω πως η μελέτη αυτή έγινε μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους και παρουσιάστηκε ως ε, ερευνητική διατριβή και θα προσπαθήσω να τα συνοψίσω όλα σε μερικές διαφάνειες. Like Ah, no, it's upwards actually. Okay. So, um, so the content of the, of the presentation. Λοιπόν, θα παρουσιάσω πρώτα το ίδιο το project, τους στόχους της ε, διατριβής, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όπως επίσης και το πεδίο. Μετά θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της μελέτης από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Πρώτα απ' όλα τα αποτελέσματα της ανάλυσης των αναφορών που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και δεύτερον τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, βελτιώσει το επίπεδο πρόσβαση στη δικαιοσύνη και έχουμε και τις συστάσεις οι οποίες διατυπώνονται στην έκθεση βασιζόμενοι στην έρευνα που έγινε. Να σας πω πως η μελέτη είχε δύο βασικούς στόχους. Καταρχήν, το να κατανοήσουμε για ποιο λόγο οι πολίτες έχουν στραφεί στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και προσπαθούν μέσω Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, αποκτήσουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ανάμεσα σε άλλα θέματα είναι τα νομικά, τα δικανικά, τα πρακτικά ζητήματα όπου τους οδηγούν σε αυτό και να σας πω πως Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, κοινωνικοί λόγοι, ιστορικοί λόγοι και πολλές φορές και πολιτικοί λόγοι. Το δεύτερο θέμα της μελέτης έχει να κάνει με την αξιολόγηση του κατά πόσο σχετικής είναι οι αναφορές και πώς χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί και εργαλεία που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να βελτιώσουν το επίπεδο πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών σε δικαιοσύνη. Δύο λόγια και για τη μεθοδολογία, την οποία χρησιμοποιήσαμε για να κλείσουμε το θέμα αυτό. Καταρχήν, το project ολόκληρο έγινε σε τρεις φάσεις. Το πρώτο στάδιο ήταν να ορίσουμε το πεδίο εφαρμογής της έρευνας, η πρώτη φάση είχε να κάνει με το τι αποτελεί αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και για το σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι κάναμε τρία βήματα. Το πρώτο βήμα ήταν το να εντοπίσουμε τις αναφορές όπως υποβάλλονται μέσω της πύλης και μέσω του καταλόγου 3 και μετά να κάνουμε μια απογραφή αυτών των αναφορών και να τις κατηγοριοποιήσουμε. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθω αργότερα. Και τέλος, επιλέξαμε αναφορές για να τις αναλύσουμε σε βάθος. Μετά, στη δεύτερη φάση, κάναμε την ερευνητική εργασία. Αυτή έτρεχε παράλληλα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιήσαμε ένα δείγμα οκτώ κρατών μελών, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετωνία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία και Σλοβακία και στόχος των, εθνικών, των ερευνών σε εθνικό επίπεδο ήταν τριπλός. Καταρχήν, να δούμε αν τα θέματα που προκύπτουν στις αναφορές ε, όντως ε, είναι σημαντικά για τα κράτη-μέλη στο δείγμα. Δεύτερον, μια καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων αυτών και επίσης να εντοπίσουμε τους παράγοντες οι οποίοι κρύβονται πίσω από αυτά τα ζητήματα. Και τρίτον, να λάβουμε ε, πληροφορίες για τις βέλτιστες ε, πρακτικές και προτάσεις για δυνητικές βελτιώσεις που θα μπορούσαμε να φέρουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ε, στο θέμα της πρόσβασης δικαιοσύνης στην έρευνα που κάναμε ε, ε, στο εθνικό επίπεδο ήταν έρευνα στα χαρτιά αλλά παράλληλα ε, κάναμε και κάποιες συνεντεύξεις με τους κομβικούς εμπλεκόμενους στα κράτη-μέλη. Οπότε είχαμε νομικούς, δικαστικούς, μη καπαόμικρον και σε κάποιες περιπτώσεις και τις εθνικές αρχές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η έρευνά μας βασίστηκε κυρίως επίσης σε έρευνα ε, στα χαρτιά με κάποιες ε, ε, συνεντεύξεις έτσι ώστε να ορίσουμε αν υπάρχει επαρκής αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να αντιμετωπίσουμε εργαλεία και μηχανισμούς που προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας που δίνουν την αρμοδιότητα στα ευρωπαϊκά όργανα για να βελτιώσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε εθνικό επίπεδο. Και σε μια τρίτη φάση αναλύσαμε ε, όλα αυτά και συντάξαμε το, τη σχετική μελέτη. Τώρα, ορισμός του πεδίου. Είναι ένα περίπλοκο θέμα η αποτελεσματική πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη και είναι δύσκολο να οριστεί, οπότε το κάναμε κυρίως μέσω του ορισμού των διαφόρων κατηγοριών που εμπίπτουν σε, στον ορισμό της αποτελεσματικής πρόσβασης δικαιοσύνης και πρέπει να σας πω πως είναι τρεις κατηγορίες και τρεις υποκατηγορίες αυτών. Θα τα πω στα γρήγορα και θα επιστρέψω αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε θέματα που είναι ε, σημαντικά γιατί περιγράφουν την ανάλυση μας. Είναι λοιπόν η αποτελεσματική προσφυγή στο δικαστήριο, περιγραφή των εθνικών ε, συστημάτων δικαιοσύνης, τα νομικά και τα πρακτικά κολλήματα. Μια άλλη κατηγορία είναι το κόστος ε, της νομικής αρρωγής και της προσφυγής σε δικαιοσύνη και αυτό έχει να κάνει με τη νομική αρρωγή αλλά και με άλλα τέλη και χρεώσεις που έχουν να κάνουν με την παροχή νομικής αρρωγής και τρίτον είναι η πρόσβαση στη δίκη και η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων. Έχουμε λοιπόν εδώ διάφορα δικανικά θέματα όπως είναι η διάρκεια της όλης διαδικασίας και επαναλαμβάνω η επιβολή των δικαστικών αποφάσεων. Η ανάλυση των αναφορών σχετίζεται με την προσφυγή στη δικαιοσύνη, την πρόσβαση σε αυτήν και στην ανάλυση που κάναμε είδαμε ότι τα πρώτα κομμάτια του, της διατριβής δίνουν τα εξής συμπεράσματα. Για τις πρώτες κατηγορίες προέκυψαν τρία ζητήματα τα οποία προκύπτουν και στις αναφορές και που παρακολύουν από την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Καταρχήν, ο τρόπος που είναι τα οργανωμένα τα εθνικά δικαστικά συστήματα και οι επιπτώσει που έχουν αυτό για την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Πώς είναι οργανωμένα τα δικαστήρια, το γεγονός πως δεν υπάρχει δυνατότητα ε, ε, προσφυγής εναντίον πρωτοδικών αποφάσεων. Επίσης, οι συνδίκες εργασίας των δικαστών, ε, κάποιοι δικαστές οι οποίες έχουν συμβάσει περιορισμένου χρόνου, για παράδειγμα, και όλα αυτά επηρεάζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε επίπεδο απλού πολίτη. Επίσης υπάρχει μια υποκατηγορία που είναι άλλα πρακτικά εμπόδια που είναι η γεωγραφική κάλυψη των δικαστήριων, το κατά πόσο στις απομονωμένες περιοχές υπάρχουν δικαστήρια, μετάφραση για τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες, όπως επίσης και η άρνηση της αποδοχής ηλεκτρονικός υπογραφής ε, στην αλλογραφία μεταξύ ε, δικηγόρων και δικαστικού σώματος ε, που επίσης προβληματίζει κάποιους, δημιουργεί πρόβλημα για κάποιους. Επίσης υπάρχουν και άλλα, κάποια, και άλλα δικανικά εμπόδια, για παράδειγμα κάποιοι αναφερόμενοι αναφέρθηκαν σε αυτά. Για παράδειγμα, απαιτήσει ταχυδρομικής διεύθυνση στη χώρα στην οποία γίνεται η, η προσφυγή ή η δικαστική διένεξη, όπως επίσης ε, και το αποδεκτό και το παραδεκτό κάποιων ε, στοιχείων ή τεκμηρίων. Επίσης, η δεύτερη κατηγορία, το κόστος της δικαιοσύνης και της νομικής αρρωγής που πολλές φορές αποτρέπουν τους πολίτες από την προσφυγή στο δικαστήριο και αυτό έχει αναφερθεί σε αρκετές ε, περιπτώσεις. Έχουμε επίσης τα τέλη, τα δικαστικά, ε, τα χαρτόσημα και επίσης το κατά πόσο υπάρχει επιδότημα πενίας ή κάποιο άλλο είδους επίδομα ε, νομικής αρρωγής που επιτρέπει την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε συχνά, για παράδειγμα σε διασυνοριακές υποθέσεις, αλλά επίσης και στην περίπτωση ορισμού δικηγόρου ή συνηγόρου ε, ή για την εξαίρεση από τα δικαστικά τέλη. Και μία ακόμα υποκατηγορία που ήταν η προσφορά δικαστικής αρρωγής σε κάποιες ε, αναφορές, για παράδειγμα, από τους ίδιους τους ε, νομικούς. Για παράδειγμα, φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα οδήγησε σε μια ενεάμινη ε, απεργία δικηγόρων στη χώρα, η οποία ουσιαστικά ήταν εμπόδιο στην προσφυγή στη δικαιοσύνη. Ξέρω και κάποια άλλα παραδείγματα οι επιπτώσεις της, ε, των κανόνων στην εσωτερική αγορά και το πώς επηρεάζουν ε, το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος για τους δικηγόρους στην Ισπανία. Έχουμε τους καθημερινούς ε, ενάγοντες οι οποίοι πολλές φορές αναφέρονται σε θέματα επιλογής δικηγόρων ή συνηγόρων που δεν τους προσφέρθηκε ή της ε, κατάρτισης ε, και της, ε, του επαγγελματισμού του δικηγόρων οι οποίοι τους ορίστηκαν και επίσης για την επιβολή εκτέλεσης δικοστικών αποφάσεων Εκεί πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλές αναφορές. Ήταν η πλειοψηφία αυτών που αναλύθηκαν και είχαν να κάνουν την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Τώρα, δικανικές εγγυήσεις και καταπάτηση αυτών είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται στις αναφορές και κυρίως το θέμα της διαφθοράς που σε πάρα πολλές αναφορές καταγγέλθηκε και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το δικαστικό κλάδο και η έλλειψη μεροληψίας και ανεξαρτησίας των δικαστών. Και αυτό αναφέρθηκε σε πολλές ε, από τις αναφορές. Η διάρκεια των διαδικασιών είναι κάτι το οποίο σε πολλές περιπτώσεις τονίστηκε ως ζήτημα Πολύ συχνά αυτό έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις ε, στα δικαστήρια και η εκτέλεση των αποφάσεων που είναι πρόβλημα σε αριθμό ε, αναφορών γιατί δεν θα εκτελεστεί μια απόφαση σε ένα κράτος μέλος ή γιατί θα καθυστερήσει η εκτέλεση. Και κυρίως για αποφάσεις που έχουμε σε περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου αλλά επίσης και στην επιβολή των αποφάσεων του ΔΕΚ ή του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. So petition... Λοιπόν, ε, εδώ βλέπουμε πολύ καλά από τις αναφορές ποια είναι τα εμπόδια στην αποτελεσματική πρόσβαση δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Και συχνά δείχνουν αναφορές ότι είναι συστημικά τα προβλήματα στα κράτη-μέλη. Οι πολίτες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρέμβουν και να λυθούν τα προβλήματα. Άρα θα έπρεπε να καταλάβουμε τι μπορεί να κάνει ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Ποια είναι τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα για να βελτιώσουν την πρόσβαση των πολιτών στην δικαιοσύνη. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο που λέγεται αναφορά πώς το χρησιμοποιούν αυτό σε σχέση με θέματα που απτώνται της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Συχνά για θέματα ε, εσωτερικά, δηλαδή εναλλακτικά προς την δικαιοσύνη της χώρας τους, όταν θεωρεί κάποιος ε, ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη του και πρέπει να κάνει αναφορά ή ότι είναι ε, πάρα πολύ υψηλή φραγμή και τα εμπόδια για να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και η πρόσβαση δεν είναι απρόσκοπτη, άρα κάνει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό ένδικων μέσων εσωτερικών ε, στη χώρα του για να αυξηθεί η πιθανότητα να δικαιωθούν. Σε μερικές περιπτώσεις επίσης χρησιμοποιούν την αναφορά γιατί υπάρχει μία έλλειψη κατανόησης, ακόμα και πώς λειτουργεί η αναφορά, για τις αξιώσεις που έχουν για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Το παραδεκτόν τώρα ε, των ε, αξιώσεων ε, και των απαιτήσεων από τη δικαιοσύνη των αναφερομένων. Αυτό είναι πιο ειδικό θέμα. Υπάρχουν κάποια κριτήρια να εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και της δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια για το πώς ερμηνεύονται αυτές οι έννοιες. Και αυτό αφήνει ένα περιθώριο στις αναφορές. Ε, πολλές φορές τέτοιες αναφορές όμως θεωρούνται παράδεκτες. Και πολλές από τις αναφορές που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, εντάσσονται στον κατάλογο 3 και δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς πριν θεωρηθούν απαράδεκτες. Αυτή τη στιγμή θεωρηθεί παραδεκτή μία αναφορά που έχει πάντα σχέση με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ακολουθεί ε, αίτημα ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιες επαφές με τα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα άλλα εργαλεία που έχει ε, στη διάθεσή του ένα θεσμικό όργανο εκτός από ε, την αναφορά τα προδικαστικά ερωτήματα και αποφάσεις. Ένα εθνικό δικαστήριο ε, παραπέμπει ένα θέμα στο ευρωπαϊκό για να ρωτήσει κάτι προδικαστικά. Αυτός ο μηχανισμός έχει πολλά ωφέλη. Πρώτον, εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία και ε, εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου εθαρρύνει εθνικές μεταρρυθμίσεις ε, στα συστήματα της δικαιοσύνης όπου δεν ε, ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και επίσης είναι και ένα μέσον για τους πολίτες να θέσουν υπόψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διάφορα προβλήματα συμμόρφωσης. Γιατί ενώπιον ενός εθνικού δικαστηρίου αν το ζητήσουν από τον Εθνικό Δικαστή είναι στη διακριτική του ευχαίρεια αν θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή όχι για να ρωτήσει κάτι προδικαστικά. Μπορεί να το κάνει λοιπόν και ο πολίτη. Το πρόβλημα είναι ότι ε, δεν γίνεται μεγάλη χρήση αυτή τη δυνατότητα προδικαστική απόφαση, γιατί ο κόσμο δεν τα γνωρίζει αυτά τα θέματα και δεν καταλαβαίνει και το μηχανισμό. Επίσης, αυτό παρατείνει και τις εθνικές ε, διαδικασίες που είναι προβληματικές ας πω στη διάρκεια από μόνες τους στη δικαιοσύνη Επίσης υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στα δικαστήρια και δικαιοδοσίες κάθε χώρα. Υπάρχουν και άλλα μέσα που έχουν στη δυνατότητά τους τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Υπάρχουν κάποια ένδικα μέσα που έχουν ε, υιοθετηθεί ε, για την καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη ε, για την νομική αρρωγή, για ε, ε, εξοδικαστικό μηχανισμό επίλυσης και διαδικτυακό. Αυτά είναι στο αστικό δίκαιο αλλά και στο ποινικό για την οδηγία για τη μετάφραση και τη διερμηνία, οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, πρόσβαση σε νομική αρρωγή και το τεκμήριο της αθωότητας. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ένδικα μέσα που διαθέτουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να μπορούν να δρουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης άλλο σημαντικό στοιχείο εδώ διότι μπορεί να βελτιώσουν μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει διάφορους μηχανισμούς προς την κατεύθυνση αυτή για να ενισχύσει και να προωθήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όπως είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα, οι ε, μηχανισμοί ε, προετοιμασίας και έγκρισης για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και ταμεία τα επενδυτικά. Και τέλος, υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα, ένα φάσμα ε, προγραμμάτων και πρωτοβουλειών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να ενισχυθούν ε, τα δίκτυα, ιστοσελίδες, ε, οι πύλες διαδικτυακές για την ε, αφύπνιση των πολιτών και την συνειδητοποίησή τους για την καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, συστήματα νομικής αρρωγής κλπ. Υπάρχει η διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, e-justice, η, η Ευρώπη σας. Ε, και υπάρχουν και ad hoc ε, ε, δυνατότητες χρηματοδότησης για διάφορες πλατφόρμες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χρηματοδοτεί τέτοια έργα. λοιπόν, και κάποιες άλλες πλατφόρμες που υπάρχουν μπορούν να προωθήσουν τους εναλλακτικού μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, όπως είναι το Solvit, ας πούμε, ή αντίστοιχα. Βάσει λοιπόν αυτών των πορισμάτων και ευρημάτων και για τις αναφορές και για τα εργαλεία που έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουμε προχωρήσει σε κάποιες συστάσεις και για τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να αντιμετωπιστούν τα θέματα που θέτουν αφορές, όπως είναι η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης. Αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε και τις υποδομές στα κράτη-μέλη, ας πούμε και υλικέ υποδομέ, τα δικαστήρια, τα κτίρια και να έχουν καλύτερε συνθήκε εργασία και υποδοχή ε, των πολιτών στα δικαστήρια. Ένα ουσιαστικό στοιχείο ε, είναι η μηχανογράφηση ε, και η χρήση αυτών των τεχνολογιών για να ε, διευκολύνεται η διεκπαιρέωση των υποθέσεων. Επίσης, η καλύτερη κατάρτιση για να βελτιωθεί η ποιότητα και η συνοχή των δικαστικών αποφάσεων. Οι δραστηριότητες επίσης αύξηση συνειδητοποίηση του πληθυσμού και προώθηση ε, εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών για να ε, σταματήσει ή να μειωθεί αυτή η καθυστέρηση που σωρεύεται στα δικαστήρια των υποθέσεων. Έχουμε προχωρήσει αυτές τις συστάσεις για τα κράτη-μέλη και μπορούν αυτές οι συστάσεις να υποστηριχθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της επιβολής ε, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο ε, δια των προδικαστικών αποφάσεων, όπως σας είπα, ε, να προχωρήσει και με διαδικασίες επί παραβάση να βεβαιώνεται ότι με σωστό τρόπο μεταφέρεται στο Εθνικό Δίκαιο Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και εφαρμόζεται. Επίσης, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει ε, τις μεταρρυθμίσεις δικαιοσύνης, ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα από τα διευθυντικά ταμεία που το υποστηρίζει αυτό που ανέφερα προηγουμένω. Και οικονομικά μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με κάποια εργαλεία πληροφορική ε, και υποδομέ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και τα διευθυντικά ταμεία και τα επενδυτικά. Υπάρχουν οι μηχανισμοί παρακολούθηση και ελέγχου επίση που μπορούν να βοηθήσουν το βαθμολόγιο ε, επίσης είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός ε, για ε, να βλέπουμε ενδεικτικά πώς προχωρούν και προοδεύουν τα κράτη-μέλη. Άλλες δραστηριότητες είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποστηριχθεί η προσπάθεια που γίνεται και τα κείμενα δίκτυα. Επίσης ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, τα οποία απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί στις διάφορες ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες που σας ανέφερα προηγουμένως. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι η αναφορά έχει αποδειχθεί πολύ σημαντικό εργαλείο για να θέτει υπόψη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων τα κακό κείμενα και τα προβλήματα και όπου δεν μπορούν να δράσουν μέσω μιας αναφοράς ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν μια ολόκληρη γκάμα, μια παλέτα δυνατοτήτων για να προχωρήσουν και να βοηθήσουν ε, την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ και αν έχετε ερωτήσει τη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ η μελέτη αυτή ανατέθηκε από το τμήμα πολιτικής ΣΥ. Την έχουμε συζητήσει πολύ. Εκ μέρους των Πρασίνων ε, ήρθε το έτοιμο για να κάνουμε αυτή τη μελέτη. Σας διαβεβαιώ ότι θα τη διαβάσουμε και ότι το ενδιαφέρον το που θα εκδηλώσει τα μέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ. Να ζητήσω από την Κομισιόν να πάρει τον λόγο για τα όσα μόλις ε, ακούσαμε. Έχουμε τη Λίντα Ζάβο. Δεν είμαι Λίντα Ζάβο, είμαι ο Αριστοτέλης Γαβριλιάδης, γιατί η συναδελφός μου είναι άρρωστη, οπότε την αντικαθιστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα εγώ διέτρεξα πολύ γρήγορα τη μελέτη πριν από την συνεδρίαση. Τη θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Χαίρομαι που η, το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας αφορά πρωτοβουλίες τη Κομισιόν, ειδικότερα το βαθμολόγιο της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γνωρίζετε. Θέλω να τονίσω ένα πράγμα ε, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ιδιαίτερα να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνης τους. Αυτό φυσικά δεν ενδιαφέρει άμεσα τη δική σας επιτροπή, την Επιτροπή Αναφορών. Εσά ενδιαφέρεστε περισσότερο για τα ατομικά δικαιώματα. Είναι όμως εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο αυτό εμείς παράγουμε το βαθμολόγιο της δικαιοσύνης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εκθέσεις κατά χώρα. Ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη που υπάρχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη, οι εκθέσει αυτέ περιλαμβάνουν εκτενή κομμάτια όσον αφορά τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένη τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, το 2016 η Κομισιόν πρότεινε και το Συμβούλιο υιοθέτησε συστάσεις κατά χώρα σε έξι κράτη-μέλη. Για να τα αναφέρουμε είναι η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Σλοβακία. Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων δικαιοσύνη του, σε άλλα κράτη-μέλη έχουμε αιτιολογικέ σκέψει, αλλά όχι συστάσει κατά χώρα. Αναχώρα, συγγνώμη. Οι συστάσει αναχώρα μπαίνουν σε λεπτομέρειε. Για παράδειγμα, στην Κύπρο υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τα ζητήματα αφρεγγιότητας ή προβλήματα με καθυστερήσει ε, στην αστική δικονομία. Στην Πορτογαλία υπάρχουν άλλα ε, πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, οπότε οι συστάσει είναι πολύ τεχνικέ, πολύ συγκεκριμένε και συνήθω τι παρακολουθούμε πολύ στενά στη διαδικασία παρακολούθηση Φυσικά η γνώμη μα. δεν έχει τόσο μεγάλη ισχύ όσο έχει στι προγραμματικέ χώρε που αναφέρατε, στι ε, χώρε οικονομική προσαρμογή, που είναι μία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή μόνο η Ελλάδα, η Κύπρος πια δεν είναι τέτοια χώρα, ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Ιρλανδία. Αλλά ε, η απόψη μα ε, έχει ισχύ στο μνημόνιο με εκτενείς αναφορές, αλλά το αναφέρατε νομίζω και στη μελέτη σας από ό,τι είδα στα γρήγορα. Η μελέτη σας λοιπόν ε, είναι ευπρόσδεκτη. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποτελεί πιστεύω τεράστια συμβολή στο όλο ζήτημα της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή σας. Σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τη διοργανική συνεργασία για το θέμα αυτό. Με μεγάλη μου χαρά τώρα καλώ τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Κύριε Βαλέσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο και δεν θα κάνω τον καλό. Δεν, με, δεν μου αρέσει το ότι είμαστε τόσοι λίγοι. Πού είναι οι πράσινοι, πού είναι τα υπόλοιπα μέλη. Κάτι πρέπει να γίνει. Η αλήθεια είναι πως για την περισσότερη παρουσίαση δεν ήμουν εδώ, αλλά ήμουν στην Επιτροπή ΑΦΕΤ γιατί είχα και εκεί μια έκθεση, αλλά δεν μ' αρέσει το ότι είναι μόνο πέντε από εμάς εδώ. Τώρα, για την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, να σας πω ότι είναι ζωτική σημασίας για όλα, για την ανάπτυξη, τη δίκαιη ανάπτυξη, για την ευημερία των πολιτών, για την καλή διοίκηση. Όταν λοιπόν προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα θέματα τα οποία επηρεάζουν την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τα όσα μας υποβάλλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε τα θέματα που τους ανησυχούν με δίκαιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί όλοι μιλάνε για το θέμα της πρόσβασης δικαιοσύνης σε όλη την Ευρώπη. Έχω να πω μόνο το εξής. Τέτοιες μελέτες δεν είναι αυτό που χρειάζεται η Επιτροπή μας. Εμείς θέλουμε οι αναφορές να αντιμετωπίζονται εμπρόθεσμα, αποτελεσματικά και με λύσεις. Άρα λοιπόν γιατί αυτή η έρευνα βασίστηκε μόνο σε ό,τι γίνεται σε οκτω κράτη-μέλη. Εντάξει, Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, ε, Ισπανία, Σλοβακία. Γιατί δεν έχουμε καθόλου υποσημειώσεις, ελάχιστες. Γιατί είναι όλα τόσο κατηγορηματικά. Ξέρετε πως ε, όσοι διαβάσουν την έκθεση αυτή θέλουν να δουν πώς έγινε η ανάλυση των στοιχείων και πώς τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με τα θέματα που μελέτης η έρευνα ή η έκθεση θα έπρεπε να βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες, σε επιστημονικά δεδομένα και σε απόλυτα ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης. Και έχω ακόμα ένα ερώτημα. Γιατί η μελέτη αυτή έχει να κάνει με τις μη παραδεκτές αναφορές. Αν δεν είναι παραδεκτές, γιατί να ασχοληθούμε. η επιλογή των αναφορών, του δείγμα δηλαδή, έχει να κάνει και με αυτές που έχουν κλείσει, για παράδειγμα, όπου εκεί έχουμε θεωρήσει πως το θέμα έχει λήξει. Και μετά, για κάποιο λόγο τις έχουμε ξανασημεριλάβει εδώ στην έκθεση. Οπότε ποια είναι η προστιθέμενη αξία του να αναλύσουμε κάποιες κλειστές αναφορές, τις οποίες εμείς, σας επαναλαμβάνω, θεωρούμε λήξασες. Ε, κάποια ιστορική αξία. Νομίζω ότι πρέπει να βγούμε μπροστά. Και το μήκος αυτής της μελέτης δεν δικαιολογείται γιατί οι αναφέροντες εδώ δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε δυνατότητα ε, λύσης του προβλήματος και έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμπρόθεσμα να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά και η συγκεκριμένη μελέτη δεν το έκανε. Και να σας πω πως οι αναφορές αυτές εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτές για μεγάλο διάστημα, οπότε και εδώ πρέπει να σας πω ότι πραγματικά αποτύχαμε γιατί δεν δώσαμε συγκεκριμένη δράση. Ζήτησα από τη Γραμματεία να μας δώσει ένα κατάλογο των κλειστών αναφορών και των μη παραδεκτών αναφορών που είναι μέσα σε αυτή τη μελέτη και πρέπει να σας πω πως χρειάζεται εξαντλητική ε, προσπάθεια και διζητικός έλεγχος και στο ιστορικό της ε, Επιτροπής μας θα πρέπει να τα μελετήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να εξασφαλίσουμε πως αυτά, αυτές οι αναφορές δεν έχουν εξεταστεί από κάποιον άλλον. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε εμείς ε, εργασία προηγούμενων Χρειαζόμαστε μελέτες για να λειτουργεί η Επιτροπή μας, αλλά χρειάζεται να έχουμε ένα πιο κατάλληλο τρόπο προσέγγισης με μειωμένες προσθεσμίες, με ταχεία δράση. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και για την αντιμετώπιση αναφορών στο μέλλον. Δυστυχώς δεν βλέπω γιατί ε, μας βοηθάει η συγκεκριμένη μελέτη. Σας ευχαριστώ πολύ και είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε συχνά μεταξύ μας είναι το γεγονός πως οι πολίτες στρέφονται προς εμάς ως ε, ε, τελευταία λύση ή σαν τη λύση όταν δεν έχουν βρει δικαίωση σε εθνικό επίπεδο και όταν επανειλημμένα δεν έχουν ακουστεί τα αιτήματά τους σε εθνικό επίπεδο, οπότε και αυτό θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη. Πολύ ωραία. Θα δώσω τώρα το λόγο, εκτός αν κάποιος άλλος έχει να θέσει κάποιο ερώτημα, θα δώσω το λόγο και πάλι στην κυρία Γας Μασό. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας γιατί αυτά τα οκτώ κράτη-μέλη το σκεπτικό εδώ ήταν να έχουμε ένα πάνελ κρατών μελών μια επιλογή βάσει κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου ε, καταγγελιών όσον αφορά την ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ορισμένε χώρε. Μια άλλη αιτία αυτή τη επιλογή ήταν να υπάρχει μια ισορροπή ε, γεωγραφική εκπροσώπηση. Να σχηματίσουμε και μια εικόνα και των αναφορών αυτών των χωρών όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν είχαν όλες εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πάμε στη δεύτερη ερώτημα, γιατί κάποιες είναι μη παραδεκτές και γιατί κάποιες έχουν κλείσει. Όπως εξήγησα, το παραδεκτό, το σύστημα το σχετικό που ορίζει τι είναι παραδεκτό και τι όχι, αφήνει πολλές αναφορές ε, πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην άκρη. Σκοπός λοιπόν εδώ ήταν να δούμε ευρύτερα τι εργαλεία υπάρχουν διαθέσιμα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να βοηθούν του πολίτε. Γιατί αυτό είναι ο σκοπό των πολιτών όταν έρχονται να σα δουν σε μια, στην επιτροπή σα. Ε, ζητούν βοήθεια. Και ενδεχομένω, ε, αν οι ε, αναφορές δεν είναι παραδεκτές ενώπιον της Επιτροπής, ίσως να υπάρχουν λύσεις που να μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη στις χώρες τους. Σκοπός λοιπόν ήταν να καταλάβουμε ποιο ποσοστό ε, τέτοιων αναφορών πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει γίνει παραδεκτό. Σκοπός ήταν επίσης να καταλάβουμε ότι όλες οι αναφορές που υποβάλλονται εδώ δεν γίνονται παραδεκτές απαραίτητες, παρόλα αυτά θέτουν ζητήματα πρόσβαση στη δικαιοσύνη που πρέπει να εξεταστούν. Any more questions? Άλλες ερωτήσεις? Όχι. Ωραία, σας ευχαριστώ τότε. Ευχαριστούμε ολόκληρο το τμήμα πολιτική ΣΥ που πάντα φτιάχνει έτσι ενδιαφέρουσες μελέτες ε, εφόσον το, ζητήσουμε και τις χρησιμοποιούμε εμεί ως εργαλείο, ως μέσο όχι μόνο στην Επιτροπή μας. Ε, τις βλέπουν πολύ. Ε, εγώ πολύ συχνά τις στέλνω και μαζί με επιστολές που στέλνω εθνικές αρχές, ε, σε ε, αναφερόμενους ως απάντηση σε πολλοί κόσμο. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ε, εκτενώς. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλες τις προσπάθειές σας και τις ευχαριστίες μας και προς το Τμήμα Πολιτικής ΣΥ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μου λένε ότι ότι χρειάζεται να κάνουμε μία συνεδρίαση συντονιστών σε 10 λεπτά από τώρα αλλά εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε με τους συντενιστές που βρίσκονται εδώ αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε ενδεχομένως αντί για απόψε να το αναβάλουμε για την επόμενη εβδομάδα όλο αυτό ως αντίδραση στο γεγονός ότι δεν ασχοληθήκαν με κάποια ζητήματα χθε που εγώ έλειπα. Μόνο ένα συντονιστή είναι παρόν εδώ. Οπότε ας κάνουμε το εξή, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και ας δούμε πώς θα έχει η κατάσταση στις 6 παρατέταρτο, σε 10 λεπτά. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, ας κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα δούμε σε 10 λεπτά πώς θα έχει η κατάσταση. Ελάτε έγκυρα.